Uh, know the rules, which are the same, so how to ask the floor. We have two topics today, so we will uh, um, try to, to, to dedicate same amount of time. Θα προσπαθήσω να αφιερώσω ίδιο χρόνο και στα δύο θέματα, ε, δηλαδή φορολογία, καταπολέμηση ξεπλήματος χρήματος και τραπεζική ένωση. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με την ε, φορολογία και τα ζητήματα ξεπλήματος ε, χρήματος τα οποία είναι πρώτη προτεραιότητα για εμάς ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουμε και μια ειδική επιτροπή, την TAX ε, 3, την η τρίτη κατά σειρά φορολογική επιτροπή και έχουμε κάνει και μια συγκεκριμένη ε, κάποιες ε, πιο εξειδικευμένες μάλλον εξεταστικές επιτροπές. Στο νομοθετικό επίπεδο έχουμε κάνει πολλά. Έχουμε καταπολέμηση ξεπλήματος χρήματος ε, την τέταρτη, την πέμπτη οδηγία. Και τώρα έχουμε θα έλεγα τους πιο προχωρημένους κανόνες παγκοσμίω ε, για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες και τα σχετικά. Είμαστε στην φάση του τριμερούς διαλόγου για να ενισχύσουμε ακριβώ τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής ε, στο θέμα αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό έργο και για άλλα ζητήματα φορολογία, όπου δυστυχώς μέχρι στιγμή, όπου ξέρετε υπάρχει ακόμα ομοφωνία στο Συμβούλιο και παρέχουμε πολύ σημαντικές ε, γνωμοδοτήσεις για την κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων, την ψηφιακή ε, φορολογία και θα σας πούμε και τις απόψεις μας οπότε σταματάω εδώ και να δώσω τον λόγο σε έναν εκ των τον κύριο Γιάνκου από την Βουλή της Ρωμανίας. Έχετε τον λόγο αγαπητέ. Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι, τιμή για μένα να συμπροεδρεύω σε αυτή την σύνοδο σε αυτή τη συνεδρίαση. Είναι πολύ προ... μεγάλη πρόκληση το θέμα. Κατανοούμε όλοι ότι αυτές οι εξελίξεις στον κόσμο δεν μπορούν να συνεχιστούν. Δεν είναι βιώσιμες αυτές οι εξελίξεις. Αντιμετωπίζουμε, θα αντιμετωπίσουμε σκληρά προβλήματα, δύσκολα. Έχουμε τρεις βασικές κατηγορίες προβλημάτων. Πρώτα η ασφάλεια. Δεύτερο, η αλλαγή του κλίματος. Τρίτον, οι κοινωνικές ανισότητες. Άπειρα περίπλοκο το σύστημά μας. Και η ισορροπία πάρα πολύ ευαίσθητη. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την ισορροπία αυτή. Οι περισσότεροι παράγοντες είναι οι περιφερειακές συγκρούσεις, αύξηση τιμής του πετρελαίου, τρομοκρατία. Αυτά είναι αντικειμενικά προβλήματα. Υπάρχουν και υποκειμενικά όμως. Αυτά συζητούμε. Ας αλλάξουμε κάπως νοοτροπία και στάση. Ας είμαστε ρεαλιστές στην προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε σήμερα. Για δύο δεκαετίες εξετάζω το όλο θέμα. Αυτά τα φαινόμενα. Εμπεριέχουν ένα παράδοξο. Ποιο? Όσο πιο θετικέ είναι οι εξελίξει, τόσο λιγότερο αποτελεσματικέ είναι. Αυτό είναι το παράδοξο. Πώ γίνεται αυτό. κατέληξα σε, σε έναν ορισμό, σε ένα απόφθεγμα που θέλω να σας αναφέρω για να το σκεφτείτε. Το ξέπλυμα του χρήματος, λοιπόν, η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή είναι συντεταγμένες του κόσμου, του ηθικού κόσμου Ο πλούτος και το μέθος του πλούτου καθορίζουν τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου σήμερα. Και αμαυρώνεται η ηθική πτυχή. Και η ηθική ρίχνεται στην κάλαθο των αχρήστων. Και το ξέπλυμα του χρήματος και η φοροδιαφυγή θα εκδηλώνουν αυτή την ανήθικη προσέγγιση στα πράγματα. Υπάρχει ένα πασίγνωστο κείμενο Τελικά οι αδύναμοι και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κινούνται με αυτόν τον τρόπο σπαταλάνε τις δικές σου ικανότητες και χαλάνε και τους άλλους. Τα Lux Leaks, τα Swiss Leaks, τα Panama Papers, όλα αυτά τα φαινόμενα πώς να τα εξηγήσουμε. Εάν, πώς να τα αναλύσουμε αν θα βρούμε τα αιτία να δούμε πώς η κοινωνία μας χάνει τις ηθικές της αξίες. Στην προηγούμενη σύνοδο, στην προηγούμενη συνεδρίαση, μάθαμε κάποια πράγματα. Αναφερθήκαμε στους κοινωνικούς δείκτες, την απασχόληση, τα κριτήρια απασχόλησης, τις σχετικές δυσκολίες, τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους, την αιρεσιμότητα, αλλά έχουμε και παράγοντες εσωτερικούς, όπως είναι οι τράπεζες, οι πολυεθνικές, τα χρηματοπιστωτικά συστήματα οι οικονομικοί σύμβουλοι. Και αυτοί οι παράγοντες κάθε χρόνο μας επηρεάζουν. Αν εξετάζουμε μόνο τις πολυεθνικές εταιρείες, βλέπουμε 60 δισεκατομμύρια να εξαφανίζονται. Μόνο από αυτές. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τόσα προβλήματα. Ίσως να είναι ενώπιόν μας κάποιες απαντήσεις. Και θα έλεγα να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε αυτού του είδους τα ζητήματα. Θα σταματήσω εδώ. Ήθελα να σας τσιγκλίσω λιγάκι. Και θα ήθελα ο Συμπρόεδρος να κανονίσει τη σειρά των ομιλητών. Ευχαριστώ πολύ για τα σημαντικά αυτά θέματα. Ο Πίτερ Γέτσεκ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Τάξη 3. Ευχαριστώ. Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως ακούσαμε και ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά σκάνδαλα στη φορολογία, στο, στο θέμα της καταπολέμησης ε, του ξεπλήματος του χρήματος και διάφορες χώρες ε, και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μαστίζονται από, αυτές, από αυτά τα σκάνδαλα. Εμείς στην Ειδική Επιτροπή κάνουμε ακροάσεις. Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ κακές πρακτικές αλλά και συστημικές ελλείμματα και κάποιοι περιορισμοί σε ό,τι αφορά το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ξέπλυμα του χρήματος και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Η δουλειά της ε, Επιτροπής ε, Τάξε 3 και ΕΚΟΝ, της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, ε, ενισχύονται αμοιβαία. βοηθούνται, δηλαδή οι δύο επιτροπές. Στι δύο τελευταίε αναθεωρήσει τη οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλήματο του χρήματο, όπου συμμετείχα, πάντα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πίεσε για ισχυρότερα μέτρα για να καταπολεμήσουμε το ξέπλυμα του χρήματο και την ε, χρηματοδότηση τη δημοκρατία, ενώ διάφορα κράτη-μέλη ήταν απρόθυμα. Η νομοθετική μας πρόοδος πηγαίνει βαθμιαία κινείται βαθμία και επηρεάζεται από, τα, από την αποκάλυψη σκανδάλων όπως τα LuxLeaks. Ε, η εφαρμογή της οδηγίας ε, για το ξέπλυμα του χρήματος είναι τελείως ε, διαφορετική από κράτος σε κράτος και αυτό, κράτος μέρος σε κράτος μέρος δηλαδή, και αυτό μας δημιουργεί προβλήματα και ανησυχίες. Γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Είναι σημαντικό επίσης να δούμε τι θα γίνει με την ψηφιακή φορολόγηση γιατί οι σημερινοί κανόνες για τη φορολογία δεν ε, καλύπτουν τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ιδίω όσων αυτών που έχουν ψηφιακή παρουσία. Και δεν είναι δίκαιο αυτό για την ενιαία αγορά. Και γενικά η δίκαιη φορολόγηση είναι ένα από τα στοιχεία για να διευρύνουμε τα ωφέλη της παγκοσμιοποίησης και να εξαπλωθούν αυτά τα ωφέλη όσο πιο πλατιά γίνεται. Πάλι φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη είναι διστακτικά, δεν μπορούν να συμφωνήσουν επί μιας κοινής λύσης. Αυτή η συζήτηση είναι πολύ επίκαιρη, συνάδελφοι. Η δική μας Επιτροπή Τάξη 3 θα υιοθετήσει την επόμενη εβδομάδα την τελική της έκθεση. Με μεγάλη χαρά, λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γέπε Φόρτ, το ένα από τους δύο εισηγητές της Επιτροπής ε, Τάξη 3 που θα παρουσιάσει σε λίγο τα βασικά πορίσματα και τις βασικές συστάσεις της Επιτροπής Τάξε 3 στον τομέα αυτό. Επίσης, ο κ. Βαλέρ Μουταλιέ, που είναι Διευθυντής για την άμεση φορολογία της Γενικής Διεύθυνσης Ταξού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος θα σας παρουσιάσει τη, τις παλιές και τις σημερινές πρωτοβουλίες της Κομισιόν στον τομέα της φορολογίας. Ο Γενικός Διευθυντής, ο κ. Μουταλιέ, έχει το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συμπρόεδροι, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι βουλευτές, με μεγάλη χαρά είμαι εδώ ε, σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, υποστήριξή του καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής ε, θητείας. Είμαστε σε τακτική επαφή, ανταλλάξαμε ε, απόψεις με την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Ε, επίσης, η τις που έκανε οι δύο ειδικές επιτροπές, τα 3 και ΠΑΝΑ, οι οποίες, όπως αναφέρθηκε, στήριξαν την ατζέντα της Επιτροπής για μια πιο δίκαιη φορολόγηση. Επίσης, ε, τα Εθνικά Κοινοβούλια εμπλέκονται όταν γίνονται επισκέψει πρωτεύουσα, όταν γίνονται συζητήσει όπω η σημερινή. Για την Κομισιόν αυτή η άμεση επαφή είναι πολύ σημαντική. Όχι μόνο για να εξηγήσουμε τι προτάσει μα, αλλά κυρίω για να ακούσουμε τι απόψει των εθνικών βουλευτών που είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα του εκάστοτε κράτου μέλου. Από την αρχή τη ε, Κομισιόν Γιούγκερ, ο επίτροπο Μοσκοβισή έβαλε το θέμα της φορολογία πολύ ψηλά στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο. Καταφέραμε να υιοθετήσουμε 14 προτάσεις, εκ των οποίων 8 έχουν σαν σκοπό να καταπολεμήσουμε την απάτη και την ε, φορολογική ε, βελτιστοποίηση και παρόλα αυτά, παρά το πρόβλημα που έχουμε την ομοφωνία η δράση μας για να καταπολεμήσουμε την απάτη και την φορολογική βελτιστοποίηση και την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης ε, γυρίζει γύρω από τρεις άξονες κυρίως. Ο πρώτος είναι αυτός της φορολογικής διαφάνειας. Καταργήσαμε το τραπεζικό απόρριτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικεύσαμε τις αυτόματες ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Σήμερα οι φορολογικές αρχές ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες απαραίτητες για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, για τις φορολογικές συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων και κρατών, για τους φόρους που πλήρωσαν οι εταιρείε χώρα ανα χώρα και για τα σχήματα ε, φορολογικής βελτιστοποίησης που έχουν φτιάξει διάφοροι φορολογικοί σύμβουλοι, τράπεζες, ε, και τα διάφορα γραφεία των δικηγόρων. Είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά να εφαρμοστούν πάρα αυτά στα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να δούμε όλα τα ωφέλη που περιμένουμε. Έχουμε, όταν έχουμε καλύτερε πληροφορίε, κάθε κράτο μέλο μπορεί να εφαρμόσει τι δικέ του φορολογικέ επιλογέ σε όλου του πολίτε του και κατοικού. Η φορολογική διαφάνεια όμω περνάει μέσα από μια ενισχυμένη συνεργασία και διάλογο με τι τρίτε χώρε για τι δικέ του φορολογικέ ε, πρακτικέ. Ε, αντιμετωπίσαμε αυτό το πρόβλημα με έναν ευρωπαϊκό κατάλογο ε, που δημιουργήθηκε το 2017 ε, για χώρες που δεν συνεργάζονται και που θα αναθεωρηθεί από τους Υπουργούς Οικονομικών τον επόμενο μήνα. Είναι ο δεύτερος πυλώνας της δράσης μας. Είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε τη φορολογική συνεργασία σε διεθνές επίπεδο. Έχουμε μια εταιρική σχέση στενή με τον ΩΣΑ ακριβώ γι' αυτό, γιατί τα πρότυπα τα οποία αναπτύσσονται στον ΩΣΑ θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, να έχουν ευρεία γεωγραφική κάλυψη, γιατί μόνο αυτή μπορεί να εξασφαλίσει την δικαιοσύνη. Αυτά τα ίδια πρότυπα εφάρμοσε η Ένωση το 2016 για να καταπολεμήσει την επιθετική, τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό μέσω της οδηγίας για αυτό το θέμα. Με βάση την πρόταση του Μαρτίου που κάναμε το 2018, θέλουμε να θεωρήσουμε τώρα τους κανόνες για τη φορολόγηση των κερδών των επιχειρήσεων και να απαντήσουμε στο δύσκολο ερώτημα της φορολόγηση των κερδών σε μια οικονομία που είναι όλο και πιο περισσότερο ψηφιοποιημένη. Η τρίτη, ο τρίτος πυλώνας είναι ο εξυγχρονισμό της ε, φορολογικής, ε, των κανόνων της φορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΦΠΑ δηλαδή, καταρχήν με την πρόταση που κάναμε για το οριστικό καθεστώς ΦΠΑ που θα μπορούσε να θέσει τέρμα στην ε, διαφυγή 58 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η κοινή ενωπημένη βάση φορολογίας εταιριών είναι ένα project για το οποίο θα σας μιλήσουν οι εισηγητές σε λίγο και που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να λειτουργούν στην χώρα. Η τρίτη πρόταση είναι να υπάρχουμε ένα υπάρχει ένας προσωρινός φόρος για τις ψηφιακές πλατφόρμες εν αναμονή ε, παγκόσμιας λύσης. Εδώ και μήνες τώρα έχουμε αυτές τις προτάσεις ε, στο τραπέζι του Συμβουλίου, αλλά δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος. Και εδώ βλέπουμε τα όρια που έχουμε λόγω του κανόνα της ομοφωνίας. Για να καταλήξω, αυτό το, αυτός ο περιορισμός είναι κάτι που προσπαθεί να καταπολεμήσει η Κομισιόν όταν ξεκίνησε μια συζήτηση ε, για το πέρασμα από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία μέσω της, της λεγόμενης πασαρέλας, του κανόνα για την πασαρέλα, για το πέρασμα δηλαδή. Θέλουμε να επιταχύνουμε το, τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων έτσι, για απαραίτητα ντοσιέ που είναι σημαντικά για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της, απάτης, φορολογικής απάτης λαμβάνοντας υπόψη ε, τον έλεγχο των Εθνικών Κοινοβουλίων, μια και το εγγυάται η συνθήκη. Θέλω λοιπόν να συμμετάσχετε σε αυτή τη συζήτηση, να συνεισφέρετε απόλυτα, ούτως ώστε να δούμε τις δικές σας απόψεις από τα κράτη-μέλη. Κύριοι συμπρόεδροι, κύριοι βουλευτές και ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Στη διάθεσή σας είμαι για να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ πολύ και δίνω πάλι την ε, προεδρία στον ε, Ροπέρτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχουμε τον ε, εισηγητή της πρότασης για την ψηφιακή φορολόγηση, τον κύριο Νταρίους Ροζάτη από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε μια πολιτική δήλωση. Το κοινοβούλιο αυτό παίρνει την υποχρέωσή του για την καταπολέμηση της ε, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και του ξεπλήματος χρήματος πάρα πολύ σοβαρά. Και βεβαίως όλα αυτά ήταν πολύ ψηλά ως προτεραιότητα από την αρχή της ηλικίας μας και με συνέπεια υποστηρίξαμε τις διάφορες νομοθετικές προτάσεις της ε, Κομισιόν. Όπως έχει αναφερθεί έχουμε εγκρίνει μια σειρά νομοθετημάτων που αφορούν τις αναφορές αναχώρα για φορολογικά ζητήματα μεταξύ κρατών μελών ε, που έχει γίνει εντωμεταξύ αυτόματη και υποχρεωτική έχουμε στηρίξει νομοθετήματα που έχουν ως αποτέλεσμα την καλύτερη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε φορολογικά ζητήματα και επίσης είμαστε πολύ ενεργοί στην εφαρμογή της οδηγίας κατά του ξεπλήματος χρήματος ε, και χρηματοδότησης της ε, τρομοκρατίας τα τελευταία χρόνια. Τούτων λεχθέντων Οφείλω να πω, τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμα τέλεια. Θα έλεγα ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις ε, στο πλαίσιο αυτό και από την δουλειά των διαφόρων επιτροπών εδώ στο Κοινοβούλιο βλέπουμε πως υπάρχουν κενά ελλείψεις ε, στο σύστημα ειδικά της καταπολέμησης του ξεπλήματος ε, χρήματος που δεν λειτουργεί επαρκώς. Μπορούμε ακόμα να πούμε ότι είναι ένα σύστημα σουρωτήρι. κάποια σκάνδαλα που ανέφερε ο σύμπροδρος ε, LuxLeaks, ε, Football Leaks, ε, Panama Papers, το σκάνδαλο CumEx και άλλα μας δείχνουν πως παρά τις προσπάθειες που έχει αναλάβει εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση το σύστημα επιτρέπει φοροδιαφυγή, φοροποφυγή και φορολογική απάτη μεγάλης κλίμακας σε τους συγκεκριμένους τομείς στους οποίους ε, βλέπουμε ότι η φορολογία δεν είναι δίκαιη και πολύ αποτελεσματική είναι η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. Οι ψηφιακές υπηρεσίες είναι ένα νέο φαινόμενο και δεν ε, αντικατοπτρίζεται επαρκώς από τους υφιστάμενους φορολογικούς κανονισμούς. Αυτό οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση και στην γρήγορη τεχνολογική αλλαγή που έδειξαν πάρα πολλούς τρόπους για την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή στον ψηφιακό κλάδο. Και όχι μόνο αυτό, αν δούμε την απόδοση του ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε πολλές δυνατότητες αποφυγής ε, των φόρων. Αλλά στην ε, ψηφιακή φορολογία έχουμε κάποιες ιδιαίτερες ε, προκλήσεις. Μια κανονική προσέγγιση στη φορολογία είναι να φορολογούνται τα έσοδα με βάση την φυσική παρουσία μιας εταιρείας, ενώ στην περίπτωση ψηφιακών εταιριών, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει φυσική παρουσία των εταιριών στα κράτη-μέλη, παρέχουν όμως ψηφιακές υπηρεσίες χωρίς να είναι παρούσες. Οπότε η Κομισιόν κατέληξε στην ιδέα ότι για να καλυφθούν αυτά τα έσοδα με, στη φορολογία για να πηγαίνει να επαρκές τμήμα στους εθνικούς ε, προϋπολογισμούς πρέπει να εισαχθεί η έννοια της ψηφιακής φορολογίας. Αυτό αντικατοπτρίζει την τρέχουσα πρακτική, όπου μια εταιρεία διαδικτυακή με βάση σε μια τρίτη χώρα παρέχει υπηρεσίες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, χωρίς, όπως είπα, να έχει φυσική παρουσία, αλλά ταυτόχρονα ε, συλλέγει εισόδημα από την πώληση αυτών των υπηρεσιών. Και μάλιστα η αξία αυτών των υπηρεσιών δημιουργείται από τους χρήστες, που είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Και κατά την άποψή μας, και εδώ πέρα συμφωνεί και η Κομισιόν και το Συμβούλιο και ο ΣΑ μάλιστα, αυτό είναι ένα σημαντικό κενό που πρέπει να καλυφθεί στο σύστημα. Ποια είναι η πρόταση λοιπόν. Η Κομισιόν έχει φέρει δύο προτάσεις για δύο νομοθετικές προτάσεις. Να συνοψίσω την πρώτη για την οποία είμαι εγώ εισηγητής. Είναι η πρόταση για να συσταθεί η ε, σημαντική ψηφιακή παρουσία σε ένα κράτος μέλος να αξιολογηθούν τα έσοδα τα οποία δημιουργούνται και να φορολογηθούν οι υπηρεσίες ε, αναλόγως με ένα σύστημα το οποίο θα κατανέμει τα έσοδα αυτά και αναλόγως μετά τα κέρδη ε, στα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν προτείνει ξεκάθαρα σαφή κριτήρια για να μετρηθεί η ουσιαστική ψηφιακή παρουσία. Αυτά περιλαμβάνουν τον αριθμό των χρηστών που έχουν εγγραφεί σε κάθε κράτος μέλος, τον αριθμό των επιχειρήσεων και το ύψος των εσόδων από την πώληση των ψηφιακών υπηρεσιών. Τα έσοδα αυτά μετά υπολογίζονται χρησιμοποιώντας μια λειτουργική ανάλυση που έχει χρησιμοποιηθεί Ήδη εδώ και αρκετά χρόνια, παραδείγματο χάρη ε, στον υπολογισμό των ε, ενδομηλικών ε, χρεώσεων σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά κέντρα παραγωγής και θα υπολογίσουν τον καταβλητέο φόρο. Δεν είναι ένας καινούριο φόρος, είναι φόρος εταιρικό, αλλά σε κέρδη τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν φορολογηθεί. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία γιατί από την πείρα μας γνωρίζουμε ότι ε, υπάρχει αρχή της ομοφωνίας στα φορολογικά ζητήματα οπότε επαφίεται στο Συμβούλιο η λήψη της απόφασης οπότε θέλουμε να σας ζητήσουμε αγαπητοί συνάδελφοι να στηρίξετε αυτή την πρωτοβουλία να πιέσετε το Συμβούλιο να λάβει μια σκληρή στάση σε αυτά τα θέματα έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη να μην στερούνται τα έσοδα αυτά από τους προϋπολογισμούς, από τις ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά αντιθέτως οι εθνικοί προϋπολογισμοί να στηρίζονται από την δίκαιη και αποτελεσματική πρωτοβουλία, ε, φορολογία, των ψηφιακών υπηρεσιών. Σας ευχαριστώ. Και τώρα συνεισηγητής για τελική έκθεση της ειδική Επιτροπής Tax 3 για Κόφορντ, της Ομάδας Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ. Η φοροδιαφυγή και η φορολογική απάτη είναι τεράστιο πρόβλημα, όπως ξέρετε, στην Ευρώπη. Μέχρι ένα 3 ευρώ το χρόνο κοστίζει εντολή για την Ειδική Επιτροπή για τα οικονομικά κλίματα, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή υιοθετήθηκε 1η Μαρτίου 2018, θητεία εντολή ενό έτου Εδραζόμεθα επί των εργασία άλλων δύο επιτροπών και μια συνεργατική επιτροπή που ασχολήθηκε με διάφορε μορφέ ε, φορολογικών απατών και οικονομικών εγκλημάτων. Ξεκίνησε εργασία με το σκάνδαλο LuxLeaks το 2014, όπω θυμόσαστε, σε αυτή τη θητεία που απέδειξε ότι κάποια κράτη-μέλη συστηματικά προσέφεραν ειδικέ συμφωνίε φορολογικέ στι πολυεθνικέ εταιρείε, επιτρέποντα στι πολυεθνικέ να μειώσουν τεχνητά ε, πολύ χαμηλά το φόρο, φορολογικό συντελεστή. Οπότε μετακυλίστηκε η φορολόγηση από τα κράτη-μέλη που είχαν υψηλότερη φορολόγηση. Αυτέ ήταν συμφωνίε που συνήπτονται με ε, συγκεκριμένε εταιρείε, ενώ ο κανονικό φορολογικό συντελεστή για τι άλλε εταιρείε παρέμεινε υψηλό χρειάστηκε ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σε ταχεία συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου, το σκάνδαλο LuxLeaks δεν μπορεί να επαναληφθεί. Τα κάτι μελη θα πρέπει να ενημερώνουν το ένα το άλλο για τις φορολογικές αποφάσεις. Μεγάλο επίτευγμα. Ασχοληθήκαμε και με τα Panama Papers, Swiss Leaks, Danske Bank, Pilatus Bank, ABLB, πολλά και ένα σύστημα μεγάλο ξεπλήματο χρήματο και πολλά θέματα. Να συνοψίσω ένα πεντάλεπτο είναι δύσκολο. Τι θα κάνω. Θα σε πιστήσω την προσοχή σε κάποια συμπεράσματα που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για του εθνικού βουλευτέ. Πρώτον, τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω δεν συνεργάζονται αρκετά καλά, γρήγορα, αρκετά γρήγορα, αρκετά συστηματικά. Από το LuxLeaks στο COMEX και Danske Bank στα Panama Papers είδαμε ότι τα κράτη-μέλη και αρχές των κρατών μελών δεν συνεργάζονται. Αυτό κοστίζει στα κράτη-μέλη δισεκατομμύρια σε απώλεια φόρων και σε απάτες φορολογικές. Το σκάνδαλο X, Φερρυπίν, εκλάπησαν τουλάχιστον 55 δισεκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα των φορολογουμένων που είχαν ήδη πληρωθεί στα ταμεία των κρατών μελών. Το 2012 οι γερμανικές αρχές κατάσχεσαν το master plan που περιέγραφε πώς άλλα κράτη-μέλη θα ήταν στόχος από εκείνου που διέπρα, διέπραταν αυτή την απάτη. Αυτά τα κράτη-μέλη όμως δεν προειδοποιήθηκαν και η απάτη συνεχίστηκε επί πολλά έτη μετά. Άλλο παράδειγμα από τη χώρα μου. Το σκάνδαλο Danske Bank. Πάνω από 200 δισεκατομμύρια ευρώ ξεπλήθηκαν από υποκαταστήματα της Danske Bank στην Εστονία. Οι αρχές, υποπτικές της Δανίας και της Εστονίας επανειλημμένα τσακώθηκαν περί δικαιοδοσίας και περί ευθύνης. Και αυτό οφειλόταν σαν ακριβή διατύπωση στην νομοθεσία Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Αλλά ήταν και αποτέλεσμα τη έλλειψη οποιασδήποτε μορφή συντονισμένου μηχανισμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω για επίλυση αυτών των θεμάτων. Η νομοθεσία κατά του ξεπλήματο χρήματο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω γνωρίζετε, έχει τη μορφή οδηγιών και όχι κανονισμών. Αυτό τι σημαίνει, ότι εφαρμόζονται ποικιλοτρόπω, διαφορετικά σε κάθε κράτο μέλο και τα βλέπουμε τα αποτελέσματα καμιά φορά. Έχουμε μια αγορά και ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίου, αλλά έχουμε 28 διαφορετικά συστήματα εποπτεία όσον αφορά τι τράπεζε, μετακίνηση κεφαλαίων κλπ. Οπότε είναι περίπλοκο το σύστημα με πολλά κενά και κρυφές γωνίες και το, τα εκμεταλλεύονται αυτά οι εγκληματίε και απαταιώνε. Δεν είναι μόνο διοικητικό πρόβλημα, πρακτικό πρόβλημα. Συμπεράναμε ότι είναι και παράβαση των συνθήκων που υποχρεώνει η συνθήκη τα κράτη-μέλη να συνεργάζονται πιστά και ειλικρινά μεταξύ τους. Δεύτερον, η μυστικότητα και οι απαιτήσει περιομοφώνιας. Το Συμβούλιο παραμένει ε, ένας λήθος που μπλοκάρει την καταπολέμηση φοροδιαφυγής, φοροποφυγής και χρηματοστικών εγκληματών όπως η οδηγία για, ε, για τη φορολόγηση των καταθέσεων. Όταν προτάθηκε το 1989 πριν από 25 χρόνια, πέρασαν 25 χρόνια μέχρι να υιοθετηθεί, ήταν ήδη απερχαιωμένος ο κανονισμός και έτσι τελικά ανακλήθηκε τον επόμενο χρόνο. Αυτό λόγω απαιτήσεων περιομοφωνίας. Όμως η οδηγία μόνο σου ζητούσε διαμήρωση πληροφοριών μεταξύ κρατών μέλων για την καταπολέμηση φοροαποφυγή. Παρ' όλα αυτά, χρειαζόταν ομοφωνία για να εγκριθεί. Αυτό είναι επιβλαβέ κατά την άποψή μου. Οφείλεται στην επικίνδυνο συνδυασμό μυστικότητε, ανωνυμία που εφαρμόζεται και στο Συμβούλιο και στι ομάδε εργασία του Συμβουλίου. Το εντόπισε αυτό και ο συνήγορο του πολίτη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ιδεολογικοί κανόνε για τη φορολογία των επιχειρήσεων και εκεί συζητούνται τα θέματα φορολόγηση των εταιριών και λαμβάνονται οι δέουσε αποφάσει. Γι' αυτό ζητήσαμε αύξηση διαφανεία τη εργασία του Συμβουλίου και των ομάδων εργασία του Συμβουλίου. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λογοδοτούν για τι δράσει του στο Συμβούλιο και στο πώ ψηφίζουν. Αυτό τονίστηκε ιδιαίτερα και στον έλεγχο πλευρά του Κοινοβουλίου των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που ουσιαστικά ο έλεγχο είναι αρμοδιότητα των Εθνικών Κοινοβουλίων, ο έλεγχο των κυβερνήσεων. Λοιπόν, μια συμβουλή, αν είχα να δώσω στου συναδέλφου των Εθνικών Κοινοβουλίων, και έχετε υπόψη μου ότι και εγώ ήμουν μέλο του Κοινοβουλίου τη Δανία από το 1998 μέχρι το 2014. Ποια είναι η συμβουλή μου, λοιπόν. Ψάξτε τι κάνει η κυβέρνησή σα, τι οδηγίε δίνει στου δημόσιου υπαλλήλου να λένε και να κάνουν στι ομάδε του Συμβουλίου, να λογοδοτούν οι εθνικέ κυβέρνησει αυτά που κάνουν και να μην παραμένουν εντό και κλεισμένων θυρών στο Συμβούλιο οι εργασίε. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Ολοκληρώνουμε τι εργασίε όσον αφορά έκθεση στην ειδική μα επιτροπή. Θα ψηφιστεί αυτή η έκθεση την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου, στην Επιτροπή και ένα μήνα αργότερα στο Κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια. Παρά τι σημαντικέ βελτιώσει, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη παραμένουν ανεπαρκή για να σταματήσουν και να διώξουν διασυνοριακέ οικονομικέ απάτε και κλίματα. Πολύ συχνά αποκαλύπτονται υποθέσει όχι από τι αρχέ των κρατών μελών, αλλά από πληροφοριοδότε, ερευνητέ, δημοσιογράφου ή ακόμα και από τι αρχέ των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό πρέπει να διορθωθεί γρήγορα. Αν θέλουμε πραγματικά να προστατεύσουμε τα κράτη-μέλη, να προστατεύσουμε τα μία των κρατών μελών να ξαναποκτήσουμε κυριαρχία στον αφορά τα φορολογικά θέματα, να σταματήσει το χρηματοστικό έγκλημα, όπω το ξύπνα χρήματο και οι φορολογικέ απάτε. Χρειαζόμαστε πολύ καλύτερη συνεργασία επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα θα βγει στην έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Hans Mikkelbach από τη γερμανική Bundestag, ε, μέλος της Επιτροπής Οικονομικών. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η φοροδιαφυγή, η καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος και τα ζητήματα φορολόγησης της ε, ψηφιακής οικονομίας μας απασχολούν και στα εθνικά κοινοβούλια. Για την Επιτροπή Οικονομικών της Γερμανικής Βουλής μπορώ να πω ότι στα θέματα αυτά έχουμε ήδη κάνει αρκετά. Γνωρίζουμε ότι η Γερμανία μπορεί να έχει μια ισχυρή οικονομία και αυτό αποτελεί έναν ε, σημαντικό παράγοντα και φοροδιαφυγής. Έχουμε πάνω από 30.000 τέτοιες περιπτώσεις που διαπιστώνονται κάθε χρόνο, οι οποίες ερευνώνται εντατικά από τις ε, αρχές. Βεβαίως το ξέπλυμα του χρήματος ε, είναι μια πολύ σοβαρή απειλή σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απειλή για το δημοκρατικό κράτος δικαίου γιατί κατά κανόνα από πίσω βρίσκεται το καρκίνωμα του οργανωμένου εγκλήματος, το ξέπλυμα χρήματος και το οργανωμένο έγκλημα ε, πρέπει να ε, αντιληφθούμε ότι πηγαίνουν μαζί ε, γι' αυτό ακριβώς ε, υπάρχουν ε, συνεχείς ανακαλύψεις και απορούμε με την ευρηματικότητα των δραστών και το ύψος επίσης των χρημάτων που ξεπλένονται. Έχουμε την σχετική οδηγία, την οποία αφού εφαρμόσαμε την Τετάρτη αναμένουμε και την Πέμπτη οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος και θεωρώ ότι η στενή συνεργασία των αρμοδίων αρχών ε, των κρατών μελών έχει πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά όπως είπα η διεθνής ε, συνεργασία στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, να αφαιρθώ λίγο σύντομα στα κράτη-μέλη Ε, τα οποία θα πρέπει να δούμε στο θέμα της ε, φοροαποφυγής. Ε, το μόνο κράτος μέλος το οποίο έχει υπογράψει τέτοιες συμφωνίες με κάποιες πολυεθνικές χωρίς καμία προϋπόθεση είναι ε, κράτη-μέλη τα οποία τελικά πλουτίζουν εις βάρος των υπολείπων. Γι' αυτό εδώ πέρα χαιρετίζουμε την πρόταση για μια ενιαία φορολογική βάση των επιχειρήσεων. Είτε ένας ελάχιστος συντελεστής είτε και κοινοί συντελεστές ε, θεωρώ ότι είναι καλά βήματα. Χαιρετίζω επίσης ότι εν ώψη της ε, φορολόγησης της ε, ψηφιακής οικονομίας ε, θα πρέπει να βρεθεί μια βιώσιμη λύση με στόχο να υπάρξει και μια διεθνής συνεννόηση. Εμείς θα προτιμούσαμε το πλαίσιο του ΟΟΣΑ, το οποίο και σε άλλες περιπτώσεις όπως τα BEPS έχει αποδειχθεί πολύ αποδοτικό. Και καλό θα ήταν κάποια κράτη-μέλη της ε, κοινότητας ε, εν τω μεταξύ ε, να ξεκινούσαν από την πορεία αλλά να μην κάνουν μονομερείς κινήσεις γιατί έτσι αποδυναμώνεται η διαπραγματευτική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να κινηθούμε και να δράσουμε από κοινού στην ε, Ευρώπη. Ε, ειδικά προς το συμφέρον των ε, επιχειρήσεών μας, οι οποίες παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε περιοχές εκτός των μεγάλων Μητροπόλεων, όσον αφορά και την παροχή υπηρεσιών και θέσεων εργασίας και κατάρτισης. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι για την πρωτοβουλία αυτή του ΟΣΑ. Τι μας φαίνεται αφίβολο το εάν είναι σωστή η πρωτοβουλία της Κομισιόν. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί. Κάτι άλλο θα ήθελα να ξεκαθαρίσω τέλος. Οποιαδήποτε προσπάθεια με τον ψηφιακό φόρο ή άλλον φόρο άμεσα ή έμεσα να δημιουργήσει μια φορολογική αρχή στην ε, φορολογική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το οποίο θα απορρίψουμε εμείς ως ε, τσέντεου τσέσου. Πρόκειται για ζήτημα εθνικής κυριαρχίας η φορολογία και προνόμιο του κάθε κοινοβουλίου το οποίο είναι αρμόδιο για τα δημόσια οικονομικά. Αυτό το λέω και όσον αφορά και τα όσα ακούγονται για κατάργηση της αρχής της ομοφωνίας στα φορολογικά ζητήματα. Η κατάργηση της αρχής της ομοφωνίας ε, δεν απαιτείται κατά την απόψή μας. Ήδη σήμερα ο μηχανισμός της ενισχυμένης συνεργασίας παρέχει αρκετή ευελιξία και ήδη υπάρχουν οι ε, συζητήσεις. Η κριτική της ε, Κομισιόν που επιζητεί να θέσει τους ε, φόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μας λέει ότι την εμποδίζει η αρχή της ομοφωνίας είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Πολύ περισσότερο θεωρώ ότι Αυτά τα οποία έχει πει η Κομισιόν είναι έκφραση μιας ε, νοοτροπίας συγκεντρωτικής, ένας ε, συγκεντρωτισμός ο οποίος ε, δεν βοηθά στην εμβάθυνση της κοινότητας, αντιθέτως μπορεί να δημιουργήσει νέα χάσματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ για τα σημεία που αναφέρατε. Υπάρχει η νομική βάση για τη φορολογία, υπάρχει και η πασαρέλα, η λεγόμενη ρήτρα γέφυρα που υπάρχει μάλιστα και στη συνθήκη. Άρα δεν συμφωνούμε όλοι με τι απόψει αυτέ. Θα δώσω τώρα το, την προεδρία στον κύριο Ιάνκου. Έχει κλείσει ο κατάλογο των μιλητών. Θα ήθελα να τηρήσετε το χρόνο σας, που είναι δύο λεπτά. Πέντε είναι οι ομιλητές. Θέλετε κι εσείς να μιλήσετε. Θέλετε τρία λεπτά. Αν χρειαστεί θα σας δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο. Ξεκινάμε. Η κυρία Μαριάννε Μίκο από την Εστονία είναι η πρώτη ομιλήτρια. Αγαπητοί συνάδελφοι, η, το ξέπλυμα του χρήματος είναι ένα διεθνές έγκλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, στην νομοθεσία δηλαδή, και να υπάρχει ισχυρή νομοθεσία μεταξύ των κρατών μελών. Η επιθεώρηση των οικονομικών στην Εστονία εντόπισε το πρόβλημα της Danske Bank. Χρειάζεται όμως ένα διεθνές πλαίσιο για να βοηθηθούμε και πρέπει να επιμεριστούμε τους κινδύνους γιατί σήμερα τα πράγματα είναι πολύ ασαφή. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχουν τα προνόμια να ερευνούν οι αρχές, αλλά σήμερα εμφανίζονται νέα ρίσκα γιατί αλλάζουν μορφή οι απάτες. Οι εστονικές αρχές έκαναν μια χαρτογράφηση για να δούμε πώς μπορούμε να καταστήσουμε πιο αποτελεσματική τη μάχη μας. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Εστονικό Κοινοβούλιο έχουμε νομοθεσία για να μπλοκάρουμε τις απάτε. Έχουμε ε, δυνατότητα παρατήρησης, ενισχυμένη δυνατότητα παρατήρησης από πλευράς των αρχών. Το βασικό είναι να καταλάβουμε τους νέους κινδύνους που αναφύονται Γι' αυτό κάνουμε νέα αξιολόγηση στο Υπουργείο Οικονομικών και είναι σαφές ότι θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ορισμός της φορολογικής απάτης, να τον ξαναδούμε αυτόν τον ορισμό. Σήμερα κάποιες πράξεις δεν θεωρούνται εγκλήματα, ενώ πρέπει να ξαναδούμε την έννοια της φορολογικής απάτης. Όταν, ας πούμε, ένα τρίτο κράτος δρά και εξαπατά τον ευρωπαϊκό ας πούμε προϋπολογισμό. Προφανώς θα πρέπει να τονίσουμε την ε, ευρωπαϊκή συνεργασία για να φρενάρουμε τις νέες ε, απάτες. Εξοικονομήσαμε και 10 δευτερόλεπτα. Χάρη στην ταχύτητά σας. Ο κύριος Γεράσιμος Βαλαούρας από την Ελλάδα. Μικρόφωνο παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ τα χαρτιά και η ενημέρωση που έχουμε είναι για τρία λεπτά αλλά το ξεπερνάω γιατί θα μου δώσετε πέντε. Ε, θα ήθελα να επικεντρώσω την ομιλία μου στα θέματα φοροαπάτης, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής που αποτελούν ένα μεγάλο σκάνδαλο κατά των πολιτών και των δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαράδεκτο ότι είτε το σύστημα φορολογικού ελέγχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι διάδεικτο και μετά από τόσα χρόνια δεν κάνουμε τα αυτονόητα είτε όταν τα κράτη-μέλη γνωρίζουν τέτοιες σκανδαλώδεις περιπτώσεις δεν κάνουν τίποτα με σκοπό την προστασία των τραπεζών και των μεγάλων εταιριών τους. Τα θέματα της φοροαπάτης είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση που απαιτείται πολύ στενότερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την δημιουργία των απαραίτητων μηχανισμών. Άρα και σε αυτή την περίπτωση χρειαζόμαστε ε, περισσότερη Ευρώπη και όχι επιστροφή σε λύσεις που βασίζονται στα κράτη-μέλη μόνο. Τόσο στο σκάνδαλο με την Google, Amazon και Starbucks και τις λοιπές εταιρείε, όσο και τα σκάνδαλα φοροδιαφυγής και πολυετούς φορολογικής απάτη CAMEX και CAMCAM, τα οποία έχουν κοστίσει παρακαλώ τουλάχιστον 55 δισεκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία, επιβορύνοντας τους εντύμους και τους συνεπείς φορολογούμενους ουσιαστικά ροκανίζοντας την εμπιστοσύνη του απλού πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτός νιώθει ότι υπάρχει έλλειψη ισονομίας και στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή η κατάσταση συνεχίζεται ακόμη και σήμερα παρά τα όποια πρόστιμα έχουν οριστεί. Και μοιράζουμε αυτό το αίσθημα αδικίας κύριε Πρόεδρε και σας ρωτάω γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει τα γιγαντιαία κλίμα της φορολογικής απάτης μεγάλων εταιριών και τραπεζών σε βάρος των δημόσιων ταμείων και των συνεπών φορολογουμένων. Χρειαζόμαστε φυσικά ευρωπαϊκές λύσεις που βασίζονται στην ευάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δικαιότερους και διαφανέστερους όρους. Πρωτοβουλίες όπως αυτή η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κόμμου για κοινέ έρευνε και ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης είναι καλοδεχούμενος και πρέπει να προχωρήσουν. Τελειώνοντας, Ας δουλέψουμε λοιπόν για να δημιουργηθούν οι ευρωπαϊκοί εκείνοι θεσμοί συνεργασίας και αυστηρού ελέγχου που θα κλείσουν τα κενά που αξιοποιούν αυτοί που φοροδιαφεύγουν ή φοροαποφεύγουν. Προ αυτή την κατεύθυνση δεδομένων των σχετικών ψηφισμάτων και του Ευρωκοινοβούλου, θα ήθελα κύριε Γουαλτιέρη, προσωπικά σε εσά να σα παρακαλέσω να ενισχύσετε σύμφωνα με τις αρχές σας και με το κύριο σας να υπάρχει σύντομα ένα συγκεκριμένο οδικός χάρτης προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you very You are... Ευχαριστώ. Σεβαστήκα τα τρία λεπτά. Και τώρα η κυρία Περβάνς Μπερέσα, Γαλλίδα Ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους τους ε, συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια που είναι παρόντες. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε μαζί και να μιλάμε μαζί για ένα τέτοιο θέμα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν και διστάμενες απόψεις. Το θέμα της ε, κυριαρχίας για φορολογικά θέματα μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με διαφορετικούς τρόπους. Θυμάμαι κάποια από τα σκάνδαλα τα οποία χρωμάτισαν την ε, επικαιρότητά μας και τις ε, εργασίες της τάξε 3. Βλέπουμε, ας πούμε, το σκάνδαλο QMEX. Ε, μία εθνική νομοθεσία επέτρεψε αυτές τις υπερβολές. Αλλά όμως οι επιπτώσεις ξεπερνούν κατά πολύ το εθνικό επίπεδο. Είναι σαφές ότι η εθνική κυριαρχία δεν μπορεί να βρει λύσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όταν βλέπουμε τις πηγές διαφυγής και φόρο-αποφυγής, δεν ξέρω πού πρέπει να βρούμε τις λύσεις. Εγώ θα πρέπει να στείλω τρία μηνύματα, πιστεύω. Καταρχάς, είμαι εντυπωσιασμένη, κατάπληκτη από το γεγονός ότι συχνά στα κράτη-μέλη υπάρχει ένας υπερθεματισμός, ειδικά σκεφτείτε την πρωτοβουλία Γαλλίας-Γερμανίας, σε ό,τι αφορά την φορολόγηση της ψηφιακής παρουσίας. Κάναμε μία γαλλογερμανική πρωτοβουλία. Αυτό ε, μας επέτρεψε να επιταχύνουμε την δράση μας. Ε, η Κομισιόν είχε βάλει και αυτή μία πρόταση στο τραπέζι και για την φορολογία των επιχειρήσεων. Η ίδια ιστορία είναι. Με κάποιους ευρωβουλευτές ε, είχαμε αυτό το όνειρο να δουλέψουμε περισσότερο με τους εθνικούς βουλευτές, με τους ομολόγους μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε μία αντίληψη που υπάρχει στο Συμβούλιο και που μας φαίνεται αντιπαραγωγική συχνά. Για, μιλάμε για την άποψη του τι είναι φορολογική, φορολογική κυριαρχία στον 21ο αιώνα. Επίσης, τρίτο μήνυμα, το θέμα του ξεπλήματος του χρήματος. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ. Είναι και αυτό μια φορολογική απάτη. Αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι και οι εθνικές αρχές, αλλά και οι ευρωπαϊκές αρχές, οι οποίες παρεμβαίνουν και κάνουν τις έρευνες ε, σε περιπτώσεις ξεπλήματος χρήματος, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα φορολογικά δεδομένα που έχουν συλλεγεί. Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει μια ρογμή στο μηχανισμό μας εδώ, πολύ ε, σοβαρή ρογμή που θα πρέπει να ξεπεράσουμε. Στα πλαίσια επίσης του τριμερούς διαλόγου που κάναμε για, με τις εποπτικές αρχές, θέλουμε υπό την αιγίδα των Ευρωπαϊκών Τραπεζικών Αρχών να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το ξέπλυμα του χρήματος. Μαρνίξ Ράι από την Πολωνία. Έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Βελτιέρη, κύριε Συμπρόεδρε, εδώ είμαι. Φαν στα γερμανικά. Φων είναι, γερμαν... είναι φαν στα ολλανδικά. Φων είναι γερμανικό. Λοιπόν, θα είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα, να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα εντυπωσιακό ιστορικό τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την ε, καταπολέμηση της αποφυγής ε, της φορολογίας και της φορολογικής ε, απάτης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ότι ο ΣΑ δημιούργησε το πρόγραμμα BEPS και η Ευρωπαϊκή Ένωση κινήθηκε αρκετά γρήγορα ώστε να πάρει αυτό το πρόγραμμα και να το μετατρέψει σε δίκαιο από ε, προαιρετικές ε, διατάξεις ε, με τις σχετικές οδηγίες. Μετά λοιπόν, το θέμα είναι ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει να το εφαρμόσουν. Και το επόμενο ερώτημα είναι εάν θα λειτουργήσουν όλα αυτά. Δηλαδή η νομοθεσία και οι κανόνες είναι το ένα, αλλά σε τελική ανάλυση οι πολίτες ε, θα μας κρίνουν από την ε, επιτυχία μας, από το αν κάτι λειτουργεί ή όχι. Και για να λειτουργήσουν αυτοί οι περίπλοκοι κανόνες, οι φορολογικές αρχές στα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν την ικανότητα να τους ε, εφαρμόζουν, να τους παρακολουθούν και να συνεργάζονται σε διασυνοριακή βασική. Ε, έχω κάποιες πολύ σοβαρές επιφυλάξεις. Ε, πιστεύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστέ. Και με βάση ποια αντικειμενικά στοιχεία και αριθμούς ε, συγκρίνουμε και πώς βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Γιατί η ικανότητα των φορολογικών αρχών δεν είναι παντού η ίδια όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των κανόνων. Το δεύτερο είναι ότι η ανταλλαγή πληροφοριών είναι πάρα πολύ καλή, αρκεί να ε, τις κάνουμε κάτι μετά αυτές τις πληροφορίες. Και ίσως να υπάρχουν και κάποιες ε, παρενέργειες ε, που δεν είχε συνειδητοποιήσει ο νομοθέτης ή δεν ήθελε Παραδείγματο χάρη οι φορολογικέ ε, αποφάσει. Ε, πρέπει να καθορίσουμε τώρα τι είναι αυτέ οι φορολογικέ αποφάσει, συμφωνίε δηλαδή με διάφορε εταιρείε. Και ω αποτέλεσμα όλων αυτών των ανταλλαγών πληροφοριών έχουμε περισσότερε ή λιγότερε τέτοιε φορολογικέ αποφάσει και περισσότερη ή λιγότερη ε, διαφάνεια. Σα ευχαριστώ. Κύριε φαν, έχετε δίκιο. Λοιπόν. Θα δώσω τώρα τον λόγο στην ε, Ματία ε, Μαρίζα, Ευρωβουλευτή. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Σημερίζω με διάφορα στοιχεία που ανέφερε η κυρία Μπέρες και που παρουσίασε και ο συγητής και που αφορούσαν τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή. Είναι αλήθεια ότι η φορολογική πολιτική είναι ένα θέμα εθνικής κυριαρχίας, αλλά είναι αδύνατον να δώσουμε απαντήσεις που δεν περνούν μέσω μιας βαθιά συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα σε αυτό το επίπεδο, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να βρίσκουμε δικαιολογίες για να μην δρούμε πάνω σε αυτά τα θέματα, διότι πάνω από όλα αυτά τα ζητήματα κάνουν τους πολίτες να γίνονται καχύποπτοι εναντί των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αρκετές ε, επιτροπές δημιουργήθηκαν, η TAX 1, η TAX 2, η TAX 3, σύντομα θα ψηφίσουμε και την έκθεση, έχουμε και την ε, Επιτροπή Πάνα 1 και την Πάνα 2, άρα δεν υπάρχει έλλειψη γνώσης όσον αφορά τις πρακτικές που ακολουθούνται για... και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε την αδράνεια. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα ποσά, τεράστια ποσά, ε, κέρδη που δεν φορολογούνται και λείπουν τα χρήματα από τα δημόσια ταμεία και δεν μπορούν να επενδυθούν σε δημόσιες υπηρεσίες στα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι μόνο μέσα από τη, από τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, αρχών των κρατών μελών πρέπει να περάσουμε, να θετήσουμε συγκεκριμένα μέτρα για να ανταποκριθούν σε αυτό το πρόβλημα. Είναι καλό που οι συνάδελφοι των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι εδώ παρόντες σήμερα για να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε πριν είναι πάρα πολύ αργά. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος. Τίμο Χαράκα από την Φιλανδία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι πολύ καλή αυτή η συζήτηση συζητούμε τα πραγματικά θέματα, τα πραγματικά προβλήματα. Η εθνική φορολογική κυριαρχία είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε παραβίαστο, ενώ η φοροδιαφυγή είναι διεθνής. Τα μέλη της Επιτροπής ΤΑΞΕ θέλουν να λαμβάνονται ε, αποφάσει με άλλο τρόπο και όχι μόνο μέσω ομοφωνία, οι αποφάσει μεταξύ κρατών μελών. Η απέτηση για την ομοφωνία είναι κάτι πολύ σημαντικό για τις χώρες. Τα ακούσαμε αυτό. Ακούσαμε πολύ ε, ένθερμα επιχειρήματα υπέρ της φορολογικής κυριαρχίας και της κυριαρχίας των κρατών μελών σαν αφορά την κατάρτιση του προπολογισμού. Δεν, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε λοιπόν την, την ίδια προσέγγιση. Τι να κάνουμε. Ίσως ένα παράδειγμα θα ήταν ο μηχανισμός ανταλλαγής ρήπων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ενός διασυνοριακού φαινομένου όπου αντιμετωπίστηκε μέσω ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Μέσω εθνικής νομοθεσίας συλλέγεται ο φόρος. Λοιπόν, απαιτείται μια ευρωπαϊκή όμως προσέγγιση να αντιμετωπιστεί το ε, διασυνοριακό θέμα. Δεν θέλουμε να παραβιάσουμε την εθνική κυριαρχία. Όλα συμβαίνουν ευθύ εξ αρχή σε διεθνέ επίπεδο. Αυτή η συζήτηση έγινε και σε επίπεδο των ιδίων πόρων τη ευρωπαϊκή Ένωσης. Έχουμε θεσμούς, Ινστιτούτα που δημοσίευσαν σημαντικές αναλύσεις και θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε έναν φόρο ευρωπαϊκό όπως ο φόρος Τόμπιν, ένας διεθνής φόρος να θεσπιστεί ή φόρος για διεθνείς δραστηριότητες, κάτι που μπορούμε να το ονομάσουμε όπως θέλετε, όπως για τον φόρο για τις εκπομπές του διοξιδίου άνθρακα. Δηλαδή να έχουμε ένα είδος βάση διεθνή φορολογική. Και αυτή η φορολογική βάση ευρωπαϊκή θα μπορούσε να είναι αρκετά ευρεία και θα μπορούσε να είναι πηγή που θα τροφοδοτεί ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο. Ευρωπαϊκό Ταμείο βέβαια πρέπει να το συζητήσουμε, συζητήσουμε τους ε, κανόνες. Κανόνες περί κατανομής των χρημάτων. Αυτό είναι σημαντικότατο. Ε, είναι αδύνατον να βρούμε μια λύση κατά την οποία 27 χώρες κερδίζουν βάση της κλίδας κατανομής και δεν χάνει κανένας. Θα είναι σημαντικό και η πολιτική συζήτηση πάνω σε αυτό. Ελπίζω να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, σεβόμενη την επικουρικότητα βάσει της διαδικασίας ε, λήψης αποφάσεων των Ευρωπαϊκών. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστώ. Τελείωσε τα πέρα η συζήτηση. Ευχαριστώ που ήσασταν και τόσο ρεαλιστές. Κάνατε κάποιες προτάσεις. Βεβαίως ε, το παράδοξο αυτό παραμένει. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες ε, προτάσεις εδώ γιατί ακόμα και αν προτείνουμε να ενισχύσουμε την συνεργασία των ε, θεσμικών οργάνων έχουμε πέντε οδηγίες για τη φορολογική απάτη για το ξέπλυμα χρήματος και τα αποτελέσματα τα γνωρίζετε. Λοιπόν, ερωτώ τους ε, συναδέλφους εάν θέλουν να κάνουν κάποια παρέμβαση και δεν ξέρω, έχουν να απαντήσουν κάτι. Νομίζω ότι ε, είναι κάτι το οποίο είναι ακόμα εν εξελίξη. Έτσι είναι ότι δεν μπορούμε ακόμα να καταλήξουμε, αλλά Θεωρώ ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων υπογράμμισαν ότι το υπάρχον πλαίσιο είναι ανεπαρκές για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα την ε, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή και δεν συζητάμε εδώ πέρα την δημιουργία την αλλαγή αρμοδιοτήτων και τη μεταφορά τους ε, από τα κράτη-μέλη στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά παρόλα αυτά δύσκολα μπορούμε να αρνηθούμε ότι το υφιστάμενο σύστημα δεν παρέχει ε, καν τις ε, επαρκείς δίκλειες ασφαλείας για να προστατευτεί η ενιαία αγορά και βεβαίως και οι προπολογισμοί των κρατών μελών από την διάβρωση της φορολογικής βάσης και την ε, μετακίνηση των ε, κερδών. Οπότε ακολουθούμε την διαδικασία του ΩΣΑ και πηγαίνουμε και λίγο παραπέρα. Και εμείς ως Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρούμε ότι αυτό είναι απαραίτητο. Επίσης ε, θεωρώ ότι η γενικότερη συζήτηση για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί η φορολογική πολιτική σε μια ιδεώδη ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αλλά θεωρώ ότι θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στο πώς θα κλείσουμε τα παραθυράκια που ήδη έχουμε και θεωρώ ότι η τρέχουσα νομοθετική πρόταση που έχουμε, η κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων, η ψηφιακή φορολογική, ο ρόλος Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής στο ξέπλυμα χρήματος, έκθεση για την εφαρμογή της ε, πέμπτης οδηγίας είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Πρέπει λοιπόν ακριβώς να συνταχθούμε γιατί οι πόροι των δικών σας ε, των εθνικών προπολογισμών επηρεάζονται από αυτό το τεράστιο φαινόμενο. Είναι ε, κυρίως τα κράτη-μέλη τα οποία χάνουν λεφτά λόγω της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Και μετά πρέπει να γίνουν δύσκολες επιλογές μεταξύ αύξησης φόρων ή περικοπής δαπανών. Οπότε εάν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα, τα παραθυράκια στο υφιστάμενο πλαίσιο, τα οποία ξεκίνησαν για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και κατέληξαν στην διπλή μη φορολογία, το γνωρίζουμε αυτό. Λοιπόν, ε, θα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση. Εντάξει, ας αφήσουμε τώρα το αν θα πρέπει να έχουμε το ίδιο επίπεδο φορολογίας ε, και την ομοφωνία ή την ειδική πλειοψηφία. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε πρώτα απ' όλα τις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει και σας παρακαλώ να διαβάσετε και τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου για το πώς θα βελτιωθεί η κοινή φορολογική βάση των επιχειρήσεων και η ψηφιακή φορολογία γιατί αυτό πραγματικά θα βελτιώσει την ε, ικανότητά μας χωρίς να δημιουργήσει μια φορολογική ένωση. Ε, αλλά θα αποτελέσει μια σημαντική βελτίωση στην ικανότητα αντιμετώπιση ε, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγής. Οπότε σα ζητώ να συμμαχίσουμε τα Εθνικά Κοινοβούλια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό, ε, να απευθυνθούμε στι κυβερνήσει μα, να δούμε τι κάνουν οι Υπουργοί Οικονομικών όταν πάνε στο ΕΚΟΦΗΝ μην χάσουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος ε, για ένα σκάνδαλο τελικά το οποίο κανένας πολίτης δεν μπορεί να αντιληφθεί και να δικαιολογήσει ότι επιβαρύνουμε υπερβολικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι γιγάντιες εταιρείε ε, πληρώνουν ε, γελίους συντελεστές. Είναι λοιπόν, τα έλεγα, μια πανευρωπαϊκή κατάσταση ανάγκης και αυτή η συζήτηση μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε κάποια πρώτα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι πραγματικά κρίμα που ε, πρέπει να στριμώχνουμε τόσα σημαντικά θέματα και το δεύτερο όμως είναι εξίσου σημαντικό είναι η Τραπεζική Ένωση να περάσω λοιπόν απευθείας στο δεύτερο θέμα και είναι μεγάλη μας χαρά που έχουμε εδώ ως καλεσμένο για πρώτη φορά από την ε, εκλογή του τον Αντρέ τον νέο πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου και χαιρόμαστε που είστε εδώ πέρα, ο Ούλρικ Μπέκερ. Επίσης, ο Γενικός Διευθυντής ε, της Αρμόδιας ε, Γενικής Διεύθυνσης. Θα τους είχα πει να έρθουν, αλλά δεν ξέρω. Νομίζω καλύτερο είναι να ανέβουν εδώ πάνω από το να κάθονται κάτω. Λοιπόν, να πω εντωμεταξύ δύο λόγια ως εισαγωγή. όπω ίσως ξέρετε, το κοινοβούλιο αυτό έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στον τομέα των τραπεζικών κανονισμών. Έχουμε ολοκληρώσει τη δουλειά μας στο τραπεζικό πακέτο μείωσης του κινδύνου και έχουμε νομίζω συνεισφέρει στο να έχουμε ένα ισορροπημένο πακέτο, δηλαδή αφενός μείωση του κινδύνου, αλλά και κάποια στοχευμένα κίνητρα προς ε, τον υγιή δανεισμό, προς την πραγματική οικονομία και έχει εισαχθεί επίσης ε, μια σημαντική διαταξή για τα έμπρελ. Έχουμε επίσης και ε, μια δικλίδα ασφαλείας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που είναι πιο ισορροπημένη από την αρχική πρόταση και νομίζω θα έχετε την ευκαιρία να πείτε στον Ανδρέα Ρία ότι Βεβαίως ε, είμαστε σίγουροι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τις αρμοδιότητες ε, του πυλώνα 2 που καθορίζονται στο σχετικό παράρτημα θα, θα λάβουν τώρα πλήρων, πλήρως υπόψη τις απαιτήσει του πυλώνα 1 και οπωσδήποτε και στην επόμενη θητεία θα υπάρξει ένας νομοθετικός γύρος ε, για την ρύθμιση των τραπεζών. Υπάρχει πολλή δουλειά που δεν έχει γίνει και είναι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν επίσης, όπως είπαμε, αυτό το πολιτικό βήμα που έγινε όσον αφορά την δικλίδα ασφαλείας, αλλά υπάρχει ακόμα ο τρίτος πυλώνας που είναι οι κοινέ εγγυήσει ε, καταθέσεων. Ε, πάρα πολύ σημαντικό για να λειτουργήσει η Τραπεζική Ένωση και θα έλεγα ότι όταν ε, συζητούσαμε το τραπεζικό πακέτο βλέπαμε έναν φαύλο κύκλο. Δηλαδή υπάρχει η τάση πολλών κρατών μελών να διατηρούν κάποια εμπόδια όσον αφορά την πιο αποτελεσματική διαχείριση της ε, ρευστότητα και του κεφαλαίου για να μην υπάρχει κατακαιρματισμός. Από την άλλη δεν έχει ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση και η εγγύηση των καταθέσεων. Τώρα λοιπόν που έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδο στην μείωση του κινδύνου είναι η στιγμή να κινηθούμε και στα δύο αυτά στοιχεία παράλληλα και νομίζω θα έχουμε μία έντονη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον συμπρόεδρό μου, τον κύριο Γιάνκου και μετά στους υπόλοιπους. Να μην χρονοτριβήσω διότι κάποιοι θέλουν λίγο χρόνο παραπάνω. Ας ακούσουμε μέσα στους ομιλητές μας. Ανδρέα Ανδρία. Από εκεί είσαι. Καλώς ήρθες. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Γκουαλτιέρη, Πρόεδρε Γιάνκου, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα στη Διακοινοβουλευτική αυτή επιτροπή να συζητήσουμε τα προβλήματα όσον αφορά την ε, Τραπεζική Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποπτεύει τι μεγαλύτερε τράπεζε στην Ευρωζώνη. Η Τραπεζική Ένωση στην αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τη διάδραση μεταξύ εθνικών τραπεζικών αρχών και εθνικών νομοθετών. Χρειάζεται ομαλή διεπαφή. Καταρχήν, να αναφερθώ στου βασικού κινδύνου στην τραπεζικό τομέα τη Ευρωζώνη και να εντοπίσω κάποιε τομεί όπου παραμένουν πράγματα πρέπει να γίνουν για να ενισχυθεί η Τραπεζική Ένωση. Εν συγκρίση με την κατάσταση πριν την κρίση, οι τράπεζε τώρα έχουν πολύ ισχυρότερη θέση όσον αφορά τη ρευστότητα και το κεφάλαιο. Η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικών των τραπεζών βελτιώθηκε, αλλά τα κόκκινα δάνεια έχουν, είναι μεγάλα για πολλέ τράπεζε και έτσι ε, επηρεάζονται τα κέρδη του και η δανειοδότηση που μπορούν να δώσουν. Λοιπόν, έχει δώσει ένα πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για τη διαχείριση ε, των, ε, των κόκκινων δανείων και τι γίνεται με δεν θέλουν να δημιουργηθούν νέα αποθέματα από κόκκινα δάνεια. Λοιπόν, η κερδοφορία των τραπεζών αξιολογούνται. Υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικό το κόστο και να είναι πιο βιώσιμε οι τράπεζε και τα επιχειρηματικά του μοντέλα. Το περιβάλλον θα πρέπει να ευνοεί τι ε, τράπεζε Ευρωζώνη. Γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει πολιτική αβεβαιότητα, είναι μετάβλητη η χρηματοστική αγορά και οι μεταβλητέ και οι οικονομικέ συνθήκε αντιμετωπίζουν προβλήματα οι τράπεζε όσον αφορά τα συστήματα πληροφορική και την ασφάλεια. Ε, διότι προχωρά και ψηφιοποίηση. Οι τράπεζες προχωρούν στο σχεδιασμό για το Brexit, οι περισσότερες διαδικασίες ε, Οι περισσότερες τράπεζες φεύγουν από τη Βρετανία και η μετακίνηση θα ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Όσον αφορά την ε, Ευρωζώνη και τις τράπεζες εκεί, οι τράπεζε που λειτουργούν στην Ηνωμένο Βασίλειο συζητούν το θέμα τη δυνατότητα εμπορία, διαχείριση του κινδύνου και πώ θα μπορέσουν να υπάρχουν υποκαταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και θα πρέπει μέχρι το Μάρτιο του 2019 να λυθούν οι εκκρεμότητε. Προχωρήσαμε από τη δημιουργία τη Τραπεζική Ένωση πριν τέσσερα χρόνια. Δεν έχει ολοκληρωθεί η τράπεζα και είναι κατακαιρματισμένο ο τραπεζικό τομέα σε εθνικά σώνια. Πρέπει εσεί, ω νομοθέτε, ε, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο να μα βοηθήσετε να ανταποκριθούμε στι επιταγέ τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω Για, τη μείωση του κινδύνου προχωρήσαμε για να προσπάθειε να καταλήξουν στη τελική συμφωνία όσον αφορά το πακέτο τη τράπεζα. Αυτό θα είναι ακρογωνίω λίθο προ την ολοκλήρωση τη Τραπεζική Ενώσεω και θα βοηθήσει να ανοίξει ο δρόμο προ ε, ένα ευρωπαϊκό σχήμα για την εγγύηση των καταθέσεων. Παραμένουν όμω αποτελέσματα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα διαχείριση ε, σε των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών σε συνοριακό επίπεδο. Οπότε και οι συγχωριακέ συγχωνεύσει εμποδίζονται για να μπορέσουμε τελικά να αντιμετωπίσουμε τυχόν πλεονάσματα στο σύστημα. Η ομαλή λειτουργία του SSM απαιτεί μεγαλύτερο βαθμό εναρμόνιση, διότι η εφαρμογή διαφόρων κανόνων και διαδικασιών σε κάθε κράτο μέλο περιπλέκει ε, τα εποπτικά καθήκοντα και υπονομεύει και την ισοτιμία στην αγορά. Αυτό ισχύει ε, για τι σωστέ ε, αξιολογίε των τραπεζών. Οι επενδυτικέ εταιρείε, ελπίζουμε να συμφωνήσουν πριν από το τέλο τη θητεία τον Ιούνιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, τόσο ώστε η εποπτεία συστηματικών ε, ε, ε επενδυτικών ε, φορέων που μοιάζουν τράπεζε να ενταχθούν στο SSM. Είναι πολύ σημαντικό, διότι θα μετακινηθούν επενδυτικέ εταιρείε στην περιοχή τη Ευρωζώνη ε, στα πλαίσια του Brexit. Καλωσορίζουμε τη συμφωνία τη Συνόδου Κορφή του Δεκεμβρίου όσον αφορά το κοινό με δίκτυα ασφαλεία για το σύστημα διάσωση, το ενίο ταμείο διάσωση για να μπορέσει να δώσει φερεγκιότητα και ρευστότητα στι τράπεζε που κινδυνεύουν. Εξακολουθώ να μα δείπει ένα κοινό πλαίσιο για ρευστοποίηση των τραπεζών, ούτω ώστε να μπορούν οι διάφορε ε, τράπεζε που χρεοκοπούν να φεύγουν ομαλά από την ε, αγορά, όπω γίνεται στη ΣΥΠΑ. Τέλο, Τώρα, για την εποπτεία, για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος, δεν ανήκει αυτό στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, αλλά δείχνει τελικά η μελέτη ότι αν λειτουργούν για να λειτουργούν σωστά οι τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται πιο συντονισμένη δράση η καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος. Η Τραπεζική Ένωση ήταν επιτυχής, γίνεται πιο θεκτικό τομέα τραπεζικό, αλλά ακόμα δεν, δείχνει, δεν δίνει μια ενιαία ολοκληρωμένη αγορά εσωτερική για τι τράπεζε και διάφοροι κλειδονισμοί σε κάθε κράτος μέλος ε, οδηγούν σε μία ενίσχυση του κλειδονισμού σε διευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, πρέπει οι νομοθέτες αυτό να το φροντίσουν και να δοθεί προτεραιότητα στο πρόβλημα αυτό την επόμενη πενταετία. Ευχαριστώ, κύριε Ενρία. Ο κύριος ε, Γκερσόν. Ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θα ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησε ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη. Τα καλά νέα είναι ότι για το τραπέζι για τις τράπεζες έχουμε πετύχει συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Οποιαδήποτε συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ποτέ τέλεια, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι γιατί είναι το βήμα, απαραίτητο βήμα για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Το πακέτο αυτό αφορά και την εποπτεία των τραπεζών και την εξυγίαση των τραπεζών. Είναι ένα σημαντικό βήμα ε, προς την κατεύθυνση αυτή της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Η ρύθμιση των τραπεζών και η κρίση μας ανάγκασε να περάσουμε σε αυτό το ρυθμιστικό πακέτο ε, τραπεζών. Η κατάσταση στην αρχή της κρίσης δεν ήταν ικανοποιητική, όπως είπε ο Ανδρέα Ενρία. Έχουμε τώρα ένα τραπεζικό σύστημα που είναι πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν 10 χρόνια πριν. Τούτου λεχθέντος ε, υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Παρότι το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώνεται δραστικά τα δύο τελευταία χρόνια και είναι το λιγότερο από το 4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση πια, όλα αυτά υπάρχουν πολλές διαφορές από κράτος σε κράτος. Και η Κομισιόν έχει υποβάλει ένα πλήρες πακέτο και στο οποίο συμμετέχει και η ΕΚΤ, ούτω ώστε να μειώσουμε το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών. Στο μεταξύ, οι τραπεζικοί κανόνες είναι η βάση, αν θέλετε. Ισχύουν και για τους 27 και για τα 27 κράτη. Στην Ευρωζώνη τώρα, λόγω της διασύνδεσης με το ενιαίο νόμισμα και της διασύνδεσης τραπεζικών συστημάτων των κρατών, θεωρήσαμε ότι ήταν απαραίτητο να βασιστούμε σε αυτή τη βάση και αυτό που κάναμε στην Ευρωζώνη είναι να λειτουργούμε μαζί με τους ίδιους τραπεζικούς κανόνες, ενώ ε, τα κράτη-μέλη εκτός, Ευρωπαϊκής, ε, εκτός Ευρωζώνης λειτουργούν, είναι πιο ελεύθερα. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για να σταθεροποιήσουμε την Ευρωζώνη στην καρδιά της κρίσης. Παρ' όλα αυτά η Τραπεζική Ένωση έχει ένα εποπτικό μηχανισμό που είναι ένας καλός πρώτος πυλώνας ε, με επικεφαλή στον κύριο Ενρία. Κάνει μια θαυμάσια δουλειά ε, εποπτεύοντας τις μεγαλύτερες τράπεζες. Επίσης έχουμε το πυλώνα της ενιαίας εξυγίανσης που όπως αποδείχθηκε πριν από λίγους μήνες ε, το σύστημα εξυγείασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί. Πέρυσι φτάσαμε στο ενιαίο, ε, προοδεύσαμε για το ενιαίο backstop για την Τραπεζική Ένωση ε, και αυτό είναι καλό, αλλά υπάρχει ε, ένα πρόβλημα, ότι είναι ατελές αυτό το πλαίσιο, ατελής αυτός ο μηχανισμός. Δέκα χρόνια μετά την έναρξη των προσπαθειών για την Τραπεζική Ένωση. Ο κίνδυνος είναι ότι θα μας πιάσει η επόμενη κρίση. Θα έχουμε δηλαδή ε, ένα σπίτι ε, το οποίο δεν θα έχει ε, στέγη καλή, δεν θα είναι στεγανή, λειτουργεί όταν ο καιρός είναι καλός, αλλά όταν δεν είναι καλός ο καιρός υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την οικοδόμηση αυτού του σπιτιού, την Τραπεζική Ένωση δηλαδή. Γι' αυτό καλωσορίζουμε τα πρόσφατα αποτελέσματα, γιατί σημειώθηκε πρόοδο στα βασικά στοιχεία της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Ε, δηλαδή το backstop ε, με το ενιαίο ταμείο για την εξυγίανση. Αυτό δείχνει και την θέληση των κρατών μελών για πρώτη φορά μετά από χρόνια να σκεφτούν θετικά πώς θα συνεργαστούν δηλαδή προς ε, ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Τώρα, ποια είναι τα πιο αρνητικά στοιχεία που δεν έχουν γίνει ακόμα, που είναι ανεπίλητα, ούτω ώστε να υπάρξει αυτό το κατάλληλο πλαίσιο που θέλουμε. Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Όχι μόνο στον τρόπο που χρησιμοποιούν τα διάφορα μέτρα που υπάρχουν, αλλά και στο ποια είναι ε, τα βασικά στοιχεία ας πούμε, αυτού του οικοδομήματος για να έχουμε μια σταθερή Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Οι αλλαγές ε, που έχουν γίνει ε, λόγω της συμφωνίας αυτής πλαίσιο ε, έχουμε σημαντικές αλλαγές και έχουμε μια προθεσμία μέχρι την, τον Ιούνιο ε, για να συμφωνήσουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Αλλά είναι μικρό αυτό το χρονικό παράθυρο. Εμείς θα συνεχίσουμε να συζητάμε τα ανοιχτά θέματα, το backstop, τα τεχνικά θέματα, τις διατάξεις για τη ρευστότητα των τραπεζών και τις διατάξεις για την εξυγίανσή τους. Επίσης, Έχουμε ένα επίπεδο, μια ομάδα υψηλού επίπεδου, ε, το οποίο ε, η ομάδα αυτή θα επιληφθεί του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων, με σεβασμό βεβαίως των προνομίων όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και του Κοινοβουλίου, αλλά και της Κομισιόν. Έχουμε την αίσθηση ότι επήγει το πράγμα, γιατί κανένα δεν ξέρει πότε θα έρθει η επόμενη κρίση, αλλά το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει και άλλη κρίση. Αν δείτε τι συνέβη στο παρελθόν, βλέπετε στατιστικά ότι οι κρίσεις ε, τα τελευταία 50 χρόνια έχουν τάσει να εμφανίζονται μεγαλύτερη συχνότητα. Ε, σε ό,τι αφορά τα, τη μόχλευση των δανείων σε άλλες περιοχές του κόσμου, ε, ο κίνδυνο δημιουργείται εκτός του τραπεζικού συστήματος. το τραπεζικό σύστημα γενικά το έχουμε στεγανοποίησει. να δεν είναι πολύ εκτεθειμένο στην εξωτερική, στις αλλά συχνά οι κίνδυνοι μεταναστεύουν αλλού, εκτός του τραπεζικού συστήματος. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Για το έντις, η λειτουργία, για ένα η... λογική για ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγύηση των καταθέσεων στην Ευρώπη και κυρίως στην Ευρωζώνη θα πρέπει να έχει δύο, βασικές, ε, δύο βασικούς πυλώνες ε, στεναρότητα και συνέπεια στεναρότητα γιατί η Τραπεζική Ένωση θα πρέπει να μπορεί να αντέχει ε, ασύμετρα, συστημικά και μη ε, σοκ και συνέπεια γιατί η αρχιτεκτονική της Τραπεζικής Ένωσης θα πρέπει να εξασφαλίζει ισότητα και να ελέγχουμε τη ε, δυνατότητα και να υπάρχει και ευθύνη μάλλον να λαμβάνονται συλλογικά οι αποφάσεις με βάση τους δύο πρώτους πυλώνες. Φυσικά οι μεταρρυθμίσεις ε, θα ενισχύσουν την στεναρότητα της, ε, του τραπεζικού συστήματος στα πλαίσια του, της ΟΝΕ. Αλλά δεν θα συνεχίσω πέρα από αυτό, αυτά, από αυτά που σας είπα. Θα σταματήσω εδώ. Ο κύριος Ιάνκου. Ναι, ξεκινήσουμε. Τελείω. Έκλεισε ο κατάλογο των ομιλητών. Λοιπόν, από του ομιλητέ ε, του πάνελ αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει ένα μηχανισμό εγγυήσεων αλλά ε, δεν είναι ολοκληρωμένο. Υπάρχουν πολλέ διαφορέ μεταξύ χωρών. Λοιπόν, θα δώσω τον λόγο τώρα στου ομιλητέ. Ξεκινάμε με τον κύριο Αλμπέρτο Μπαρνάη από την Ιταλία. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ και τους άλλους ομιλητές. Μία σύντομη παρατήρηση. Ε, υπόθηκε ότι η μείωση των κινδύνων ανοίγει τον δρόμο για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και τον διαμερισμό του κινδύνου. Δηλαδή είναι δύο φάσεις. Πρώτα μειώνουμε τον κίνδυνο και μετά περνάμε στην εγγύηση. Από την Ιταλική σκοπιά ε, φαίνεται σαν να προτείνουμε το εξή πρόγραμμα. Πρώτα μειώνουμε εμεί τον κίνδυνό μας και μετά μοιραζόμαστε ε, τους δικούς σας κινδύνους. Κάτι το οποίο μας φαίνεται κάπως άδικο. Δηλαδή, έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Ειδικά προς τον κύριο Ενερία. Αναφέρθηκε ότι πρέπει να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Τι είναι με τον ρόλο των στοιχείων ενεργητικού επίπεδου 2 και επίπεδου 3 στον προπολογισμό στον ισολογισμό των Ευρωπαϊκών Τραπεζών δεν τα αναφέρατε, αλλά συχνά αναφέρονται στην συζήτηση ως μια δυνητική απειλή στην ε, οικονομική σταθερότητα της Ευρωζώνης. Αυτή είναι μια ερώτηση. Και έχω και μια άλλη γρήγορη παρατήρηση. Αναφέρατε την χαμηλή κερδοφορία του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος. Θα έπρεπε να θυμόμαστε ίσως ότι τα χαμηλά επιτόκια και το χαμηλό ευρώ πετούνται όταν ε, έρχονται οι κραδασμοί και μετά το σοκ για να διαμεριστεί ο κίνδυνος μεταξύ βορείων και νοτίων χωρών της Ευρωζώνης. Ε, υπό μια έννοια λοιπόν ε, κάτι θα έπρεπε να δαχτούμε από αυτό το διαρθρωτικό, δομικό χαρακτηριστικό της Ευρωζώνης. Σας ευχαριστώ που σεβαστήκατε και τον χρόνο. Ο κύριος Τορναρίτης από την Κύπρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να μιλήσω την ε, μητρική μου γλώσσα. Τη Τραπεζική Ένωση δεν πρέπει να παραμείνει ευσεβή πόθος και ευχολόγιο. Πρέπει να επιδειχθεί αναγκαία πολιτική βούληση και δέσμευση για επίτευξη προόδου στα πιο ουσιώδη και ευαίσθητα ζητήματα που εκκρεμούν και σχετίζονται με τη μείωση του κινδύνου και ιδιαίτερα τον επιμερισμό του ανάμεσα στους Ευρωπαίους εταίρους. Είναι αδύρυτη ανάγκη να προχωρήσουμε άμεσα σε συγκρότηση ενός κοινού δημοσιονομικού μηχανισμού προστασίας, Common Fiscal Backstop, για το ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων, ώστε να παρέχεται ίση προστασία στους καταθέτες ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Χρειάζεται να πάυσει το παράδοξο η δημοσιονομική εποπτεία και εξυγίανση να επιτελούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ η προστασία των καταθετών να παραμένει εθνική αρμοδιότητα. Προέρχομαι από μια μικρή χώρα που κατέβαλε ακριβό κόστος και τίμημα από αυτή την παραδοξότητα λόγω της οικονομικής και τραπεζικής κρίσης. Σήμερα βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση να θωρακίσουμε την, την Τραπεζική Ένωση με τους κανόνες τόσο της πειθαρχία όσο και της αλληλεγγύης. Η υιοθέτηση αυτών των μέτρων θα αποτελέσει μια τέτοια χειροπιαστή απόδειξη κοινοτικής αλληλεγγύης προς τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και τους πολίτες μας που παρά την πρόοδο που πετύχαμε αρκετοί ταλανίζονται ακόμη από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Έχουμε μπροστά μας το ορόσημο των ευρωπαϊκών εκλογών και θέλουμε να απευθυνθούμε προς τους ε, πολίτες, προς τους Ευρωπαίους πολίτες ενισχύοντας τις φιλοευρωπαϊκές τάσεις και αναχαιτίζοντας τις αντιδραστικές και συκοφαντικές δυνάμεις που πολεμούν το κοινό μας σπίτι, που πολεμούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you very much. Thank you. The first speaker... Ευχαριστώ. Hans Michelbach από τη Γερμανία. Κύριε Πρόεδρε, από την ε, δική μου τη σκοπιά Θεωρώ ότι έχουμε κάποιες ε, ουσιαστικές ε, προκλήσεις που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα εν ώψη των ευρωεκλογών. Ε, πολλά από τα συστήματα τα οποία σταθεροποιούσαν την παγκόσμια τάξη πλέον δεν λειτουργούν επαρκώς και είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια ευρωπαϊκή συνοχή. Με τον Brexit δεν ξέρουμε τελικά τι θα γίνει και η οικονομική ε, ζημία από την πολιτική οικονομικής περιχαράκωσης ε, είναι ήδη ορατή. Ο κόσμος ε, περιέρχεται σε μία αταξία χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα κάποια νέα τάξη. Και βλέπουμε ότι τα ζητήματα τις πολυμέρειες υποχωρούν. Είπα, Κίνα και Ρωσία εργάζονται προς ε, το συμφέρον της κάθε μία και σε πολλές ε, περιπτώσεις έχουμε, με παρά... έχουμε να κάνουμε με κινδύνους ε, πολύ θεμελιώδους, πολύ θεμελιώδους με και υπάρχει μια αμοιβαία ενίσχυσή τους, κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα πολύ γρήγορο τέλος ε, της δεκαετούς ε, φάσης ε, ανάπτυξης, κάτι το οποίο δεν σημαίνει βεβαίως ότι πρέπει να μας εμποδίσει στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης είναι σημαντική και αναγκαία, αλλά πρέπει να πατάει σε γερά θεμέλια και η διαδικασία μείωσης ε, του κινδύνου, ειδικά ακριβώς ε, στα κόκκινα δάνεια, είναι κάτι το οποίο έχει αποφασιστική σημασία. Και εδώ πέρα πρέπει να ληφθούν ε, φιλόδοξα μέτρα, ώστε τελικά να επιτύχουμε λύσεις οι οποίες θα είναι αποδεκτές παντού. Η πρότασή σας για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων, το ΕΔΙΣ, να αντιμετωπίζεται αφενός ε, κάπως επικριτικά στα κρατη και πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτό. Η ολοκλήρωση του λοιπόν χωρίς να αντιμετωπίσουμε επαρκώς ε, τα κόκκινα δάνεια πρώτα ε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να δεχτούμε. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να υπάρξει μια μείωσή τους για να επέλθει μια σταθερότητα γιατί ε, είναι πολλά αυτά τα οποία διακυβεύονται για την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Περβάν Μπερές λοιπόν είναι η τελευταία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους διάφορους ομιλητές που έκαναν ε, μια αποτίμηση καταστάσεως της Τραπεζικής Ενώσεως. Θα πρέπει να διατηρήσουμε την ιστορική μας μνήμη των διαφόρων υποχρεώσεων που ανελήφθησαν. Καμία φορά νομίζω ότι περιοδικά ξαναγράφουμε την ιστορία. Ξεκινήσαμε λοιπόν το σχέδιο αυτό της Τραπεζικής Ενώσεως. Είναι πάνω αυτό το σχέδιο. Τα πρώτα στάδια της Τραπεζικής Ενώσεως ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2012. θέλαμε να προχωρήσουμε με τρία πόδια, αν θέλετε. Το θέμα της εγγύησης των καταθέσεων. Είχε εξεταστεί αναλυτικά. Και ανάλογα με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται, η προσπάθεια τη μείωση του κινδύνου ε, αποκτούσε όλο και περισσότερη σημασία και ο επιμερισμός ε, του κινδύνου γινόταν ανυπέρβλητο εμπόδιο. Και βόλευε να παραμείνουν όλοι στα εθνικά του συστήματα. Όταν συναντόμαστε έτσι, τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να προσμετρήσουμε τα αντιπαραγωγικά αποτελέσματα και τα πολιτικά μηνύματα που αποστέλλονται όταν έχει αναλυφθεί μια υποχρέωση και εν ονόματι της αλληλεγγύης μάλιστα και ποτέ δεν ξεπερνάμε αυτό το βήμα να υλοποιηθεί η υποχρέωση. Επό ιδιωτικού θεσμού εξαρτάται εγγύηση καταθέσεων σε κάποια κράτη-μέλη. Δεν ξέρω τι ένομε τάξει των διαφόρων κατομέλων. Οι δημόσιε αρχέ δεν μπορούν να επιβάλλουν σε ιδιωτικού φορεί ε, δεσμεύσει. Αυτή η συζήτηση λοιπόν πρέπει να μα οδηγήσει να, σε άλλα επίπεδα, πέρα από τις τεχνικές λεπτομέρειες. Να εξετάσουμε τις πολιτικές πτυχές. Εάν οι υποχρεώσει δεν γίνονται σεβαστές και ζητούνται όλο και περισσότερε προσπάθειες, παραβιάζεται αυτή η σύμβαση, αυτή η συμφωνία και δημιουργεί απογοήτευση και αντιευρωπαϊκά συναισθήματα. Και αυτό δεν είναι προ όφελο κανένα. Ευχαριστώ. Ο κ. Μάρκο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ για την Τραπεζική Ένωση η συζήτηση συνδέεται με το θέμα του επιμερισμού των κινδύνων. Το είπε και ο κ. Μπανιάη. Είναι σημαντικό. Ο κίνδυνος ε, της πίστοσης ε, έχει μειωθεί ε, και επομένως πρέπει να δούμε και τα στοιχεία ενεργητικού δεύτερου και τρίτου επίπεδου που οδηγούν σε διαφοροποίηση στην αγορά και μπορούν να οδηγήσουν σε, χασούρα για τις συστημικές τράπεζες, σε απώλειες. Και αυτό είναι το, ο δεύτερος πυλώνας Τραπεζικής Ένωσης ε, που σημαίνει ότι σε περίπτωση κρίσης συνεισφέρουν οι καταθέτες. Επομένως, αν υπάρξουν προβλήματα και δεν έχουμε το σύστημα αγγής των καταθέσεων, θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα να διαχειριστούμε. Θα έχουμε άτομα που θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες ε, λόγω της διαδικασίας του Μπέιλιν. Σε ό,τι αφορά ε, την αξιολόγηση που γίνεται για τις α, προβληματικές πιστώσεις, πολλές χώρες έλαβαν, από το, έλαβαν ε, κρατικές ενισχύσεις, ε, μεταξύ των οποίων και η Ιταλία, αλλά η Ιταλία έχει βάλει λιγότερη ρευστότητα στο σύστημα. Στο σύστημα. Χρειαζόμαστε χρόνο γιατί και ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός δημιούργησε πολλά προβλήματα στις τράπεζες και οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν κάποιο χρόνο για να αντιδράσουν. η ε, κυρία Νουή και ο Σόιμπλε κάναν ε, διάφορες ε, συζητήσεις. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν αν συνεχίζεται στην ίδια άγουσα ή μήπως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτά τα στοιχεία, ε, να τα εντάξουμε στο μηχανισμό μας και όχι να, να απευθυνθούμε ας σε εξωτερικές δυνάμεις, κερδοσκοπικά ταμεία κτλ. Μήπως θέλει άλλος να λάβει το λόγο. Όχι. Εν τη αυτή περιπτώσει έχουμε ερωτήσεις ανησυχίες απέχουμε πολύ από τους στόχους μας. Από τον έλεγχο του κινδύνου όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα. Ο κ. Σαρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιάνκο. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις, ευχαριστώ για τα σχόλια. Καταρχάς, όσον αφορά το σχόλιο του κ. Μπανιάη, θεωρούσα σαφές ότι η πόλωση της μεταξύ μείωσης του κινδύνου και επιμερισμού αυτού ήταν κάτι επιβλαβές. Ήμασταν πολύ καλοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο να επιδιώκουμε οδικούς, να ακολουθούμε οδικούς χάρτες. Πρέπει να καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο τελικός στόχος, απότερος στόχος. Το έλεγε και ο Λιβιέ Γκέρσαν πρέπει να δούμε και όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να φτάσουμε στο στόχο. Αυτό απαιτεί παράλληλα βήματα σε όλους τους τομείς. Είναι σαφές ότι η μείωση του κινδύνου πρέπει να επιτευχθεί. Επετεύχθη σημαντική πρόοδος. Το SSM ήταν πολύ σημαντικό πλαίσιο για να επιτευχθεί η πρόοδος. Επίσης είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε και πρόοδο και στα άλλα μέτωπα. Και χρειάζεται παράλληλη πρόοδος σε δύο τομείς. Για το σύστημα εγγύσεως καταθέσεων. Καμία αντίρρηση δεν υπάρχει, πιστεύω, ότι στο τέλος της διαδρομής, μέσω του δικού χάρτη, χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγύσεως καταθέσεων. Κατά διάρκεια της κρίσεως, πιστεύω, ότι ήταν σε κάποιες φάσεις πολύ επιζήμιο το ότι εκφραζόταν ανησυχίες σε κάποιες χώρες όσον αφορά την αντοχή κάποιων συστημάτων εγγυήσεως καταθέσεων μέσω εκροής κεφαλαίων. Σε συγκεκριμένες χώρες υπήρχαν τα προβλήματα. Και έχουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να εξασφαλίζεται ε, να καλύπτονται ε, οι καταθέσεις. Αυτό το σύστημα εγγυήσεων πρέπει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να εφαρμόζεται. Αλλιώς ένα ευρώ που κατατίθεται σε μια χώρα δεν θα έχει την ίδια αξία όσο ένα ευρώ που κατατίθεται σε άλλη χώρα. Αν δεν υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή κάλυψη καταθέσεων. Ενώ αυξάνουμε τις αμοιβέ εγγυήσει μας, θα πρέπει να ελέγχουμε και τον κίνδυνο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες όσον αφορά το δίκτυο ασφαλείας στο backstop για ε, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι κάτι που κινείται προς παρόμοια κατεύθυνση. Όσον αφορά ε, για τα στοιχεία ενεργετικού επίπεδου 2 και 3, να πω δύο πράγματα. Ένα που βλέπει προς το παρελθόν και ένα προς το μέλλον. Βλέποντας τι γινόταν στο παρελθόν, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πολλέ προσπάθειες κατεβλήθησαν από το SSM σε αυτό το τομέα, κάτι που αναγνωρίστηκε πρόσφατα και στην έρευνα που έχει γίνει στην Ευρωζώνη. Έγιναν επιτόπιες, επιτόπιοι έλεγχοι, εξετάστηκαν συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια και έγιναν και δοκιμές αντοχής που ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο που ακολουθήθηκε εκεί με ιδιαίτερη μεθοδολογία για την κάλυψη ελήψεως ρευστότητας των στοιχείων ενεργητικού. Κυρίως ελέγχθηκα τράπεζες που είχαν ε, μεγάλα χαρτοφυλάκια με ε, μη ρευστά στοιχεία ενεργητικού επίπεδου 2 και 3. Όταν κοιτάμε προς το μέλλον δεν τελειώνει η ιστορία, χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια, αυξανόμενη προσπάθεια. Γιατί? διότι όσο κινόμεθα προς έξοδο από τη μη συμβατική νομισματική πολιτική που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα και εξακολουθούμε να έχουμε, είναι σαφές ότι ο κίνδυνος της αγοράς και άλλοι κίνδυνοι θα γίνονται πιο σημαντικοί. Άρα και τα διάφορα μέσα που χρησιμοποιούνται ίσως δημιουργούν προβλήματα. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πάντα σχεδίαζε εκστρατεία επιτόπιων ελέγχων για την αξιολόγηση των κινδύνων. Να δούμε τώρα για τι γινόταν στη λογιστική και τα θέματα συνετής διαχείρισης και πρόληψης και το πλαίσιο πρόληψης. Αυτό είναι κάτι που θα γίνει το 2019 και το 2020, έχει προγραμματιστεί, είναι στο πρόγραμμα εργασιών. Τώρα, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που χρειάζεται κάποιο χρόνο για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Διαφωνώ με αυτά που υπόθεται. Δηλαδή, αν δώσουν περισσότερο χρόνο για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετωμένων δανείων, βοηθούμε τι τράπεζε και τον οικονομικό τομέα και το οικονομικό σύστημα που εξυπηρετούν, αυτό το επιχείρημα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Κοιτάξτε τι εμπειρίε που έχουμε σε άλλε δικαιοδοσίε. Χώρες, οι χώρε που επλήγησαν περισσότερο όσον αφορά την κληρονομιά που αποκόμισαν σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια Αυτές ήταν οι χώρες που εξηγίαναν ταχύτερα τις τράπεζες και έφεραν τις τράπεζες σε μια κατάσταση να μπορούν να διανοδιωτούν και να είναι και κερδοφόρες. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό συνεπάγεται και δημόσια στήριξη και στήριξη του, η οποία αυτή η υποστήριξη ε, από το δημόσιο τομέα αποπληρώθηκε εγκαίρως. Η καθυστέρηση της προσαρμογής όμως εν γέννη αποκρισταλώνει καταστάσεις δυσλειτουργία των τραπεζών. έχει 50% των στοιχείων ενεργητικού που είναι μη εξυπηρετούμενα, δεν δανειοδοτεί η τράπεζα, δεν είναι επικερδής, είναι δυσλειτουργική τράπεζα, όπως αποκαλούν πολλοί. Τέλος, όσον αφορά το θέμα του BlackRock που αναφέρθηκε, απαντήσαμε σε ερωτήσεις του Γερμανικού Κοινοβουλίου διαβιβάστηκαν τον κύριο Σόιμπλε, αλλά οι ερωτήσει ήταν Γερμανού βουλευτού και υπευλήσαν και ρωτήσαν το Ευρωκοινοβούλιο πιο πρόσφατα. Πράγματι, οι σύμβουλοι του BlackRock ενεπλάκησαν στις, στα... στις δοκιμές αντοχής. Ζητήσαμε να υπάρχουν μέτρα ασφαλείας και διαχωριστικά μεταξύ των συμβούλων που εργαζόταν επί και είχαν πρόσβαση στις πληροφορίες μας μόνο επί τόπου. Να θυμηθούμε ότι για σημαντικούς θεσμικούς φορείς όταν ολοκληρωθεί εργασία δημοσιεύονται οι πληροφορίες και είναι διαθέσιμες τη πάση. Δεν υπάρχει συγκριτικό όφελος πλέον, ανταγωνιστικό όφελος για εκείνους που συμμετέχουν στην προσπάθεια. Τούτου λεχθέντος συμφωνώ. Πράγματι, πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας εξωτερικούς συμβούλους για αυτό το έργο, για αυτό στον προπολογισμό για φέτος αποφασίσαμε να εσωτερικεύσουμε αυτές τις λειτουργίες και στις οι επόμενες δοκιμές αντοχής θα γίνουν κυρίως μέσω εσωτερικών πόρων. Ευχαριστώ. Άλλος που θέλει να μιλήσει. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ γρήγορα. Συμφωνώ, όπως πάντα, με αυτά που είπε ο Ανδρέα Ρίες. Η Περβάς Περέζ καλά τα λέει. Έχει δίκιο. Πράγματι, μέχρι τώρα εργαζόμαστε βάσει το δικού χάρτη του Ολλανδικού, που συνετάχθη από το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ τον Ιούνιο 2016. Και για τη μείωση του κινδύνου και για το μερισμό του κινδύνου προχωρήσαμε. Ίσως όχι αρκετά. Αλλά όπως είπε ο Ανδρέα, φτάσαμε στο τέλος της προσέγγισης αυτές όσον αφορά το να δρέπουμε καρπούς. Ε, πρέπει να πάμε στο δεύτερο στάδιο. Η προσέγγιση σύμφωνα με την οποία χρειάζεται συμφωνία όσον αφορά το στόχο μας. Δηλαδή να έχουμε μια τραπεζική ένωση που είναι εξοπλισμένη στο να την Ευρωζώνη. Και τι συνεπάγεται αυτό. Αν ρωτήσετε τον κύριο Τρία και τον κύριο Σόλτς, ποιος είναι ο προορισμός μας, ποια θέλετε να είναι η εικόνα που θα δούμε το 2030, θα έχετε παρόμοιες απαντήσεις. Αν τους ρωτήσετε για το ταξίδι, πώς πάμε από το σημείο α στο β, ίσως να έχετε διαφορετικές απαντήσεις. Το θέμα δεν είναι ο προορισμός, το θέμα είναι το ταξίδι. Όλοι συμφωνούν βασικά ότι χρειάζεται να σταθεροποιηθεί η Ευρωζώνη όσον αφορά το τραπεζικό τομέα. Το πρόβλημα είναι πώς πάμε εκεί και τους διάφορους κινδύνους, ηθικός κινδύνος. Εξαρτάται από την τοποθέτησή σου, η άποψή σου. Αυτό είναι φυσικό. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από τη στήρα συζήτηση της μείωσης κινδύνου και του κινδύνου. Να δούμε πού θέλουμε να πάμε. Συμφωνούμε ότι αυτό θέλουμε να έχουμε. Κάποτε. Και μπορούμε να αποφασίσουμε για ποιες πτυχές μας ικανοποιούν, τι ικανοποιεί τους μεν, τους δε δυσαρεστεί, να βρούμε ε, ένα, μια συνένεση. Το θέμα είναι η σειρά που θα ακολουθήσουμε για τα βήματα. Υπάρχουν και σειρέ που είναι αδύνατο, αλληλουχίε που δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε. Χρειάζονται όλοι διαβεβαιώσει. Οι διαβεβαιώσει ποιε είναι. Ότι έχουμε μια απόφαση που έχει θεσπιστεί σε νόμο. Αυτά πρέπει να γίνουν με αυτή τη σειρά. Αυτό τώρα αποφασίζεται τι θα γίνει και με ποια σειρά. Όπως είδαμε, αν αρχίσουμε με τη μείωση του κινδύνου, εκείνοι που πιστεύουν ότι η μείωση του κινδύνου πολύ σημαντική θα θεωρήσουν ότι ποτέ δεν είναι αρκετό να φτάσουμε στον επιμερισμό του κινδύνου. Αν είχαμε ξεκινήσει με τον επιμερισμό του κινδύνου, δεν θα ήταν καλύτερη κατάσταση. Εκείνοι που ήταν υπέρ του επιμερισμού του κινδύνου έλεγαν ότι δεν είναι σημαντική μείωση του κινδύνου. Αυτό πρέπει να λύσουμε. Ελπίζω λοιπόν αυτή η ομάδα εργασία υψηλού επίπεδου θα βρει τη διέξοδο και θα ανεβάσει τη συζήτηση, το επίπεδο τη συζητήσεως βάσει των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής ε, αυτής για την Ευρωζώνη. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Ανδρέα, ότι για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, για το χρόνο αντιμετωπίσει των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αν κάναμε ένα ασφάλμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την άποψή μα, κατά την μου, είναι ότι έχει εστιαστεί πολύ σε ρυθμιστικέ λύσει που ασχολούνται με το θέμα τη ευθύνη όσον αφορά το ισοζύγιο. Σορεύοντα περισσότερε ευθύνε και παθητικό για να εξορροπήσουμε το συλλογισμό, θεωρούσαμε ότι πετυχαίνουμε το στόχο μα. Αληθεύει, αλλά είναι πολύ δαπανηρή η λύση. Άλλο τρόπο. Όχι ρυθμιστικό όσο πολύ, αλλά υποπτικό. Να εστιαστούμε στην άλλη πλευρά του ολογισμού, στην αξιολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού. Και αυτό είναι ένα τρόπο αντιμετωπίσεω των ε, μη ε, εξυπηρετούμενων δανείων ή μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων. Είναι πιο φθηνό τρόπο να το κάνουμε, γι' αυτό επικεντρωνόμαστε πάνω σε αυτό. Και με το θέμα τη κληρονομιά, αν θέλετε, των παλαιών τέτοιων μη εξυπηρετωμένων στοιχείων ε, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έχουμε αυτή την κληρονομιά, αν θέλετε, και διαφέρει από χώρα σε χώρα των κόκκινων δανείων. Εμεί πιστεύαμε ότι μπορούμε με ένα άλμα να περάσουμε τον ένα κόσμο στον άλλον. Δεν γίνεται όμω. Έχουμε θέματα παλαιών τέτοιων μη πρωτομένων δανείων που πολλούσαν ομόλογα οι τράπεζε στον παλιό καιρό στου πελάτε διατηνόμενε ότι αντιστοιχούν σε λογαριασμό ταμιευτηρίου, αποταμιεύσει. Λοιπόν, όταν όμω γίνεται το bail-in, ε, αυτό παίζει ρόλο. Οπότε η κληρονομιά μα έχει σημασία. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε τις παλιές ιστορίες, την κληρονομιά για να ξεκινήσουμε φρέσκοι. Καλύτερο, καλύτερη αυτή η προσέγγιση παρά η προσέγγιση που βασίζεται στην, αν θα συμφωνούμε επιμείωση του κινδύνου, επιμερισμού του κινδύνου. Ευχαριστώ. Να συνοψίσω. Και να απευθύνω και ένα ερώτημα προς τον κύριο Γκολτιέρη και προς τον κύριο Ανρία. Κατάλαβα ότι ε, συνοψίζοντας θα έλεγα τις σημερινές παρεμβάσεις ότι υπάρχουν δύο σημαντικά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ο ένας είναι αυτός ο εγγυητικός μηχανισμός, ο άλλος είναι η διάκριση μεταξύ χωρών, η διαφοροποίηση. Ας σας δώσω το, δεν ξέρω, ένα παράδειγμα ή μια λύση. Κάθε μέρα πληρώνουμε 1,13 δισεκατομμύρια ευρώ για ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πληρώνουμε επίσης 180 δισεκατομμύρια ευρώ για ε, τεχνολογία, προϊόντα τεχνολογίες που παράγουν ενέργεια. Φέτος ίσως 200 δισεκατομμύρια. Από πού προέρχονται αυτά τα λεφτά, από τις τράπεζες. Από πού, ποιος ε, στηρίζει αυτόν τον μηχανισμό. Οι καταναλωτές. Είναι ένας μηχανισμός επιδότησης. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να μοιραστούμε αυτές τις επιδοτήσει με τις τράπεζε, γιατί οι τράπεζε είναι τμήμα αυτή τη διαδικασία. Ίσως αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση για έναν μηχανισμό εγγύησης, γιατί από ό,τι κατάλαβα υπάρχει ένας κίνδυνος ότι οι χώρε δεν θέλουν να εμπλακούν γιατί είναι πλέον έκτημα για τι τράπεζε, αλλά σε τελική ανάλυση πληρώνουμε αυτά τα τεράστια ποσά σε καθημερινή βάση. Είναι τα μεγαλύτερα ποσά που δίνονται για την ενέργεια παγκοσμίω και την χρειαζόμαστε αυτή την τεχνολογία, την πληρώνουμε για τις επόμενες ε, δύο δεκαετίες. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ συνάδελφε για νομίζω είναι και πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και συμφωνώ και με τις ε, τελευταίες παρατηρήσεις του Ανδρέα και του Ολιβιέ θα ήθελα να φέρω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ε, συμφωνώ απολύτως με τον Ανδρέα Νερία ότι καμιά φορά ο ορισμός δηλαδή ε, όταν λέμε για την μείωση του κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και να μην βοηθά. Αυτό το οποίο συχνά μιλάμε και λέμε επιμερισμό του κινδύνου είναι ένα μέτρο μείωσης του κινδύνου γιατί αν λάβουμε υπόψη πως ήδη έχουμε μια νομική υποχρέωση, όπως έλεγε ο Ανδρέα, να δοθεί η εγγύηση για κάλυψη των καταθέσεων μέχρι τα 100.000 ευρώ. Αυτό υπάρχει ήδη, δηλαδή αποφασίζουμε μόνο για το επίπεδο αξιοπιστίας αυτής της εγγύησης και αξιοπιστία σημαίνει να καταστήσουμε λιγότερο ε, πιθανό τον κίνδυνο επέλευσης αυτού του γεγονότος. Ε, Οπότε είναι... υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του ΩΣΑ που έκανε μια προσωμείωση για το πώς ακόμα και μια πλήρης εγγύηση ε, τελείως αμοιβεοποιημένο κεφάλαιο, κατά οποίο δεν υπάρχει κανένας πρόταση, ε, σε κατάσταση κρίσης ε, τελικά θα μπορούσε να σημάνει έναν διαμερασμό των πόρων μεταξύ των κρατών μελών. Ενώ από την άλλη, αν μετρήσουμε το αποτέλεσμα που θα είχε ε, ως ένα μέτρο εμπιστοσύνης δεν σημαίνει ότι ό,τι κερδίζει ο ένας το χάνει ο άλλος. Αντιθέτως θα είχαμε ένα θετικό αποτέλεσμα συνολικά. Είναι λοιπόν καλό αυτό το οποίο είπε ο Ολιβιέ ότι δεν νομίζω κανείς να μπορεί να αμφισβητήσει τον στόχο αλλά συζητάμε την πορεία. Και νομίζω ότι η νοοτροπία που θα ήθελα εγώ να βλέπω Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να βλέπω τους Ιταλούς ε, να μιλούν για την ανάγκη της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ε, τους Γερμανούς ε, και τους Γάλλους να μιλάνε για καλύτερη αξιολόγηση των στοιχείων επίπεδου 2 και επίπεδου 3. Να υπάρχει δηλαδή μια κοινή δέσμευση για μια ισορροπία οπωσδήποτε, για την μείωση του κινδύνου, αλλά ταυτόχρονα να ολοκληρωθεί και το τραπεζικό πλαίσιο, γιατί και αυτό είναι ένα μέτρο μείωση του κινδύνου. Τώρα, για τα ιστορικά θα έλεγα δάνεια αυτά, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Χρειάζεται οπωσδήποτε μια δικλή ασφαλεία για την ροή και τη ζητηματό με ποια ταχύτητα θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την κληρονομιά δανείων. Γιατί εάν υπάρχει, παραδείγματο χάρη, ένα δάνειο με εγγύηση και ένα χωρί και πούμε ότι ε, η πιθανότητα μη πληρωμής είναι η ίδια και αν πούμε ότι οποιοδήποτε δεν είναι πιθανό να πληρώσει θα πρέπει να μηδενιστεί σε βάθος δύο χρόνων ε, δεν είναι θέμα ε, μείωσης κινδύνου μπορεί αντιθέτως να δώσει ένα περίεργο κίνητρο όσον αφορά την ε, δυνατότητα να διατηρηθούν και βιώσιμες εταιρείε. Οπότε, εδώ πέρα δεν μιλάμε για μια εξασθένηση της ε, δικλείδας ασφαλείας. Αντιθέτως και βεβαίως, εντάξει, το απόθεμα. Αυτό βεβαίω είναι κάτι το διαφορετικό και όταν εξαντληθεί θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μετά και οι κρατικέ ενισχύσει και τα σχετικά. Έχουμε λοιπόν ένα αρκετά καλό τραπεζικό πακέτο το οποίο μα δίνει ένα παράθυρο ευκαιρία και ένα αρκετά καλό κίνητρο από αυτήν την πλευρά. Ε, δηλαδή να υπάρξει ε, μια, ένα γρηγορότερο ξεκαθάρισμα του ισολογισμού των ε, τραπεζών και ένας ε, επιταχυμένος ρυθμός μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τώρα η ομάδα εργασίας υψηλού επίπεδου θα είναι πραγματικά υψηλού επίπεδου. Ελπίζουμε λοιπόν ε, το υψηλό αυτό επίπεδο να μην μας κάνει να ε, απομακρυνθούμε από τα συγκεκριμένα μέτρα για έναν οδικό χάρτη προς το σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Βεβαίω έχουμε και εμείς μια ευθύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί δεν δώσαμε τη δική μας ανάγνωση για το θέμα αυτό της εγγύησης ε, καταθέσεων και εγώ, και εγώ δεν αντιταχθήκα σε αυτό το μέτρο. Ελπίζω λοιπόν ότι ε, η επόμενη Ευρωβουλή θα μπορέσει βραχυπρόθεσμα και όχι μακροπρόθεσμα να κλείσει αυτό το κενό στο αριθμιστικό μας πλαίσιο να ολοκληρωθεί αυτό το τρίτο σκέλος και έτσι να ανοίξει τον δρόμο έτσι ώστε στον επόμενο γύρο και επανέρχομαι σε αυτό το οποίο είπε ο Ανδρέας στην αρχή να μην υπάρχουν και αυτά τα εμπόδια για την ε, τραπεζική ολοκλήρωση. Η τραπεζική ολοκλήρωση δεν σημαίνει βεβαίω ε, θα υπάρχουν τα ίδια για όλου. Ε, χρειαζόμαστε και μικρέ τράπεζε, κοινοτικέ τράπεζε κτλ. Αλλά και να υπάρξει και ένα βήμα προ τα εμπρό για την διασυνοριακή τραπεζική και θα πρέπει να σταματήσει αυτό ο βάβλο κύκλο μεταξύ κατακαιρματισμού, ολοκλήρωση Τραπεζική Ένωση και εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου. Θεωρώ λοιπόν ότι στην επόμενη θητεία θα είμαστε σε θέση να κάνουμε αυτά τα βήματα προς τα μπρος ε, εκ παραλλήλου. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε. πάρα πολύ και ελπίζω την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε να έχουμε προχωρήσει λίγο παραπέρα όσον αφορά αυτό το στοιχείο της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Να ευχαριστώ τον Ανδρέα Ανρία και τον Ολιβιέ και όλους σας και τον Συμπρόεδρο και να σας ενημερώσω πως θα έχουμε και μια μικρή δεξίωση και ένα ε, όρθιο γεύμα βλέπω εδώ πέρα στον οίκο της ευρωπαϊκής ε, ιστορίας ε, και θα μας φιλοξενήσει βεβαίως και το Ρουμανικό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να ευχαριστήσω τη γραμματεία, ευχαριστεί και τους διερμηνείς ο πρόεδρος. Καλό βράδυ λοιπόν, να περάσουμε και τα λέμε αύριο.